Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we can begin our important meeting this afternoon. Καλημέρα, συνάδελφοι. Έχουμε σημαντικό προσκεκλημένο απόψε. Καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τους λοιπούς ε, διακεκριμένους ε, προσκεκριμένους μας στην σημαντική αυτή συζήτηση για τα δύο σύμφωνα του ΟΗΕ. Έχουμε λοιπόν και εμείς αποφασίσει να ασχοληθούμε με αυτήν την διαδικασία, αφιερώνουμε χρόνο και πόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι έχουμε εδώ πέρα βουλευτές ασχολείται με αυτήν την πολύ σημαντική συνεδρίαση και βεβαίως καλωσορίζω και τους πολλούς διακεκριμένους ε, καλεσμένους μας εδώ. Και βεβαίως ε, θα έχουμε και άλλους ε, κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Η κυρία Βίξτρομ θα συνεδριάσει επίσης μια συνεδρία Αγαπητοί βουλευτές ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αγαπητέ Επίτροπε του ΟΗΕ για την ε, προστασία και τους πρόσφυγες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ορίζω επίσης και τον ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνδιοργανώνει αυτήν την συνεδρίαση. Δυστυχώς λόγω των καιρικών συνθήκων στην Σόφια η κυρία Γκοσντάνοβα πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας δεν μπόρεσε να έρθει. Ε, λυπούμαστε. Δυστυχώς κολλείεται. Η άλλη συνεδρία, όπως είπα, θα είναι υπό την προεδρία της συναδέλφου μου, της κυρίας Βίξτρομ. Σας καλωσορίζω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι στην συνεδρίαση αυτή γιατί έχουμε μία διαδικασία, είμαστε... Έχουμε εδώ πέρα 33 βουλευτές από 19 κράτη-μέλη και από την Νορβηγία, χώρα ΕΟΧ. Για εμάς αυτό αποδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των Εθνικών Κοινοβουλίων για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως είπα, από τη μεγάλη σημασία στις διαδικασίες και για τα δύο σύμφωνα αυτά του ΟΗΕ και αναγνωρίζουμε έτσι ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία να καταλήξουμε σε κάποιες αρχές και δεσμεύσεις που αφορούν την διεθνή μετανάστευση σε όλες τις, τις διαστάσεις. Κανείς δεν υποτιμά τις δυσκολίες βεβαίως και πρέπει να εμπλακούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε με μια αντιπροσωπεία υπό την Προεδρία της κυρίας Βίξτρομ στην σχετική σύνοδο κορυφής που υιοθέτησε την διακήρυξη της Νέας Υόρκης. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ λοιπόν είχε εμπλακεί ευθύς ε, εξ αρχής και συμμετείχαμε σε μια σειρά δράσεων ε, με στόχο την ενεργή εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία. Έκτοτε είχαμε διάφορες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας που αφιερώθηκαν στα παγκόσμια αυτά σύμφωνα σε συνεργασία με άλλες επιτροπές όπως η Επιτροπή Εξωτερικών και η Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσκεκλημένους μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία αγαπητοί συνάδελφοι να συναντηθούμε με συνάδελφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και με την Επιτροπή Εξωτερικών και με τον κύριο Επίτροπο για να προχωρήσουμε την διαδικασία παραπέρα σκεφτήκαμε να γίνει αυτή η συνεδρίαση για να μεγιστοποιηθεί η εμπλοκή των συναδέλφων από Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι μεγάλο τμήμα της ε, συζήτησης ε, γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Σημειώστε παρακαλώ για πρακτικούς λόγους ότι έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ιρλανδικής έχει διαρθρωθεί η συνάντηση με τρόπο απλό για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Η πρώτη συνεδρία θα συζητήσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες. Η δεύτερη θα εστιάσει στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή Ομαλή και Εφτακτή Μετανάστευση. Έχουμε λοιπόν Εμπλεκεί όλοι σε διαφορετικά επίπεδα και από διαφορετικές σκοπιές ε, και σκοπεύουμε έτσι να διαχειριστούμε την ανθρώπινη κινητικότητα ανά τον πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζουμε ένα ψήφισμα, το οποίο θα είναι έτοιμο τον Μάρτιο, όμως ε, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια συλλογική διαδικασία και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για την οικοδόμηση συνένεση. Ελπίζω λοιπόν η σημερινή συνεδρία να συνεισφέρει σε αυτό. Τέλος, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στην συνεδρίαση, στο συνέδριο του Μαρόκου αργότερα φέτο, και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεισφέρει και αυτό στις διάφορες φωνές που ακούγονται για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θετικό αυτό πνεύμα Χαίρομαι τώρα που θα δώσω τον λόγο στον συναδελφό μου, τον κύριο Κριστέα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Καλώς ήρθατε λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κλοντ ε, Μωράς, ε, ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτή τη διακοινοβουλευτική συνάντηση σήμερα και ευχαριστώ και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθαν εδώ στις Βρυξέλλες για αυτή τη συζήτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση σε βάθο με βουλευτές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει μεγάλη υποστήριξη προ τι προσπάθειε του ΟΗΕ να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη μετανάστευση και του πρόσφυγες. Παρακολουθούμε λοιπόν ε, τι διαδικασίε του Παγκοσμίου Συμφώνου από στενά, ξεκινώντα από τη Σύνοδο ε, του 2016 για του μετανάστε και του πρόσφυγε και τι διαβουλεύσει και τι δραστηριότητε απολογισμού πέρυσι. Παρακολουθούμε στενά τι διακυβερνητικέ ε, διαπραγματεύσεις που μόλις ξεκίνησαν και θα κάνουμε τη φωνή μα να ακουστεί στι διαπραγματεύσει και θα έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα υιοθετηθεί το Μάρτιο. Η μετανάστευση είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα, όπως αναφέρθηκε από το Γενικό Γραμματείο του ΟΗΕ πρόσφατα. Ο αριθμός των μεταναστών ε, υπολογίζεται στις 260 εκατομμύρια παγκοσμίω και αναμένεται να αυξηθεί διάφορα προβλήματα όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η κλιματική αλλαγή ε, και οι διάφορες εξελίξεις σε διάφορα μέρη του κόσμου θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσει σε ανθρώπου ώστε να εγκαταλείπουν τι χώρε του αναζητώντα ένα καλύτερο μέλλον. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πρόκειται να πάψει να υπάρχει. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη τη το ζήτημα αυτό. Έτσι λοιπόν απαιτείται να συνεργαστούμε ο ένας με τον άλλο ώστε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της μετανάστευσης και, της αναγκα... και τον με τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τόσο τους μεταναστές και τους πρόσφυγες όσο και τις ε, κοινωνίες φιλοξενίας, υποδοχής και τις χώρες καταγωγής. Θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες ώστε να γίνεται με τακτικό τρόπο η μετανάστευση, ώστε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ε, να μην αποτελούν το αντικείμενο εκμετάλλευσης και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκόσμια μετανάστευση. Αυτό ακριβώς προσφέρει το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Είναι η πρώτη φορά που οι κυβερνήσεις ε, κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν ένα ε, ενιαίο σύνολο κανόνων αντιμετώπιση τη μετανάστευση και του προσφυγικού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σχέδιο 0 που δημοσιεύτηκε πριν από μερικέ εβδομάδε ε, θέσπισε αρχέ και δεσμεύσει που πιστεύω θα αποτελέσουν άριστη βάση για τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις. Προσβλέπω να ακούσω τις απόψεις των ομιλητών μας και των εθνικών βουλευτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κριστέα και όπως βλέπετε συνάδελφοι, ο κύριος Κριστέα έρχεται από την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ε, αυτό αντιστοιχεί στην ολιστική μας προσέγγιση όσον αφορά αυτά τα έγγραφα. Θα παρατηρήσετε και από τους προσκεκλημένους μας και στα δύο τμήματα της Συνόδου ε, πόσο σημαντικό είναι για μα ε, που αφαιρώνουμε τόσου πολλούς πόρους σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο η κεντρική ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο, ε, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ με μεγάλη χαρά στη συνάντηση, επειδή έχει εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία και θα μας πει ποιε ήταν οι δικές του δράσει σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Κύριε Αβραμόπουλο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ για να συζητήσουμε ε, για το θέμα της έγκρισης και υιοθέτησης περί τα τέλη του έτους των Παγκοσμίων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε ε, να διευθετηθούν θέματα τα οποία αφορούν την ασφαλή ομαλή τακτική μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της διεθνούς συνεργασίας και που θα καθορίσει το κληροδότημα το οποίο θα αφήσουμε πίσω μας. Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουμε ευρύτερη κοινή κατανόηση σχετικά με το πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε όλοι μαζί με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο, αλλά και μακροπρόθεσμα, το θέμα της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Ίσως γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Νέα Υόρκη και συναντήθηκα με τον Αντώνιο Κουτιέρεθ, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Λις Χάρμπορ, την εκπρόσωπο ε, για την μετανάστευση, καθώς επίσης ε, και τον καλό μου φίλο, πρόσωπο του Υπουργείου ε, Εξωτερικών της Σλοβακίας. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τα τρία προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ενίσχυσε την συνεργασία της ε, με κεντρικές ε, χώρες στην διαδικασία της μετανάστευσης. Πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ε, παγκόσμια συνεργασία. Γιατί εξηγούμε. Πρώτον, διότι οι πολίτες μας θέλουν εμείς να διαχειριστούμε καλύτερα την μετανάστευση. Το ζητούν, το απαιτούν. Δεύτερον, διότι αυτό το θέμα δεν αποτελεί ευθύνη μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των μεμονωμένων κρατών. Είναι παγκόσμια ευθύνη. Τρίτον, διότι οπωσδήποτε οφείλουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και να είμαστε πιο έτοιμοι για το μέλλον. Πράγματι, ενδεχομένως στο μέλλον ε, θα αντιμετωπίσουμε και άλλες ε, κρίσεις ε, τέτοιου είδους, αλλά δεν πρέπει να μας βρουν απροετοίμαστους, όπως μας βρήκε η κρίση πριν από λίγα χρόνια τη στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη βρέθηκε σε μια πρωτόφαντη κατάσταση. Από ευρωπαϊκής πλευράς και προοπτικής το ζήτημα της μετανάστευσης ε, δεν έχει ακόμα λυθεί και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Για κάθε ένα από τα παγκόσμια σύμφωνα θα πρέπει να επιτύχουμε σωστή ισορροπία σαν αυτήν που προσπαθούμε εμείς να διατηρήσουμε όσον αφορά την συνολική μας ε, μεταναστευτική πολιτική. Η προσέγγιση την οποία από κοινού στην Ευρώπη έχουμε αναπτύξει τα τελευταία τρία χρόνια έχει ήδη ξεκινήσει να δίνει αποτελέσματα. Οι αφήξεις το 2017 είναι κατά 20% χαμηλότερες από ότι το 2014 πριν από την κρίση. Τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται καλύτερα. Ε, η διαχείρισή τους είναι ορθότερη. Και οπωσδήποτε ε, και οι συνθήκες ε, διαβίωσης των μεταναστών σε τρίτες χώρες, όπως την Τουρκία ας πούμε, έχουν βελτιωθεί. Επίσης, κατά 50% έχουν αυξηθεί αιτήσει ε, ασύλου ε, και έχει σε όλες τις χώρες επιταχυνθεί ε, η διαδικασία. Επίσης έχουν ληφθεί αποφάσεις για επιστροφές παρατύπων μεταναστών, έτσι ώστε να διευρυνθεί η ασφάλεια των υπολείπων. Βεβαίω, ε, βασιζόμαστε πολύ στα μελλοντικά σύμφωνα ταυτοχρόνως όμως. Η συζήτηση για τα παγκόσμια σύμφωνα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει και ευκαιρία για να αλλάξει το αφήγημα περί την μετανάστευση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το πόσο πραγματικά βασίζομαι σε εσά, στους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ε, και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια βασίζομαι σε εσά ε, για να μεταδώσετε ε, μηνύματα τα οποία θα βασίζονται όχι σε μύθους και σε μυθοπλασίες, αλλά σε πραγματικά περιστατικά και στοιχεία. Επιτρέψτε μου λοιπόν ε, να ε, μοιραστώ μαζί σας κάποια σχόλια για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το Global Compact ε, για τους πρόσφυγες, GCR. Ο αριθμός των ανθρώπων που πιθανόν να μετακινηθούν έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 65,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Βλέπουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το μεταναστευτικό έχει φτάσει πραγματικά στα άκρα. Και επομένως το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα ικανοποιητικό πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ε, θα είναι ιστορική σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βεβαίως συνδεδεμένη στην προσπάθεια να αποτρέψει ε, νέες συγκρούσεις και να επιλύσει ε, υφιστάμενες. Ε, γιατί πρέπει να σας πω ότι παρά τις προσπάθειες το να πολεμήσει κανείς τις αιτίες της μετακίνησης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, και πριν λυθούν τα προβλήματα στη Συρία ή αλλού, χρειαζόμαστε ένα μεγάλο βαθμό αλληλεγγύης και προσπάθειας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον τεράστιο αριθμό των εκτοπισμένων. Η προστιθέμενη αξία του Global Compact για τους πρόσφυγες είναι να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις έτσι ώστε συλλογικά να είμαστε σε θέση να προλάβουμε, να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τους εκτοπισμένους ανθρώπους, αυτούς που προσπαθούν να ξεφύγουν από συγκρούσεις και προβλήματα με τον τρόπο αυτό και μέσω του Παγκοσμίου Συμφώνου θα μπορέσει να γίνει καλύτερος επιμορισμός και των ε, ευθυνών, στόχο των οποίων συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μηχανισμούς αντοχής σε κρίσεις και στην Ευρώπη, αλλά οπωσδήποτε και ε, με τους εταίρους μας ε, εκτός της ε, Ευρώπης. Κατά την έννοια αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στο ύψος των δεσμεύσεών της. Το 2016 672.000 άνθρωποι έλαβαν το καθεστώς προστασίας, διεθνούς προστασίας. Το 2017 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν προστασία σε 3.082 ε, ε, ανθρώπους, κυρίως προερχόμενους από το Ιράκ και το Αφγανιστάν και τη Συρία. Ταυτοχρόνως στην Αφρική και στην ε, ε, Μέση Ανατολή υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν υποδεχθεί ε, πολύ μεγαλύτερους αριθμούς προσφύγων και βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε και τις χώρες αυτές. Κατά την έννοια αυτή η, δήλω, η διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορεί να αποτελέσει έναν καλό τρόπο βοήθειας και υποστήριξης ε, ε, χωρών ε, όπως η Τουρκία που υποδέχεται πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η διευκόλυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία με συνολικό προϋπολογισμό 3 δις ευρώ αποτελεί ένα σωστό εργαλείο έτσι ώστε από ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι θέματα υγειονομικής ε, κάλυψης, ε, κοινοοικονομικής ε, αρρωγής και ανθρωπιστικής βοήθειας ή εκπαίδευσης μπορεί λέω να αποτελέσει για όλα αυτά ένα πολύ καλό μέτρο στήριξης. Οι άνθρωποι μετακινούνται ε, προσπαθώντας να αποφύγουν τον κίνδυνο μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς. Το να βοηθήσουμε τις γειτονικές χώρες σημαίνει ότι θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους εκτοπισμένους, ώστε να μην πέσουν στα νύχια των διακινητών και έτσι ώστε να μην ξεκινήσουν μακριά και πολύ δύσκολα επικίνδυνα ταξίδια. Γίνεται προσπάθεια συντονισμού βεβαίως των χωρών οι οποίες ε, έχουν ε, ε, στο έδαφος τους πολλούς πρόσφυγες. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε τις νόμιμες διόδους για να ανακουφιστεί η πίεση σε αυτές τις χώρες. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ε, του σχεδίου μεταγκατάστασης ε, του Ιουλίου 2015 η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ε, μέσω αυτών των μέσων είχαμε μία επανεκατάσταση 27.000 προσφύγων. Θέλουμε να πάμε παραπέρα ακόμα και να επανεγκαταστήσουμε 50.000 άτομα τα επόμενα δύο χρόνια. Μέσω του Παγκόσμιου Συμφώνου περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο θα εμπλακούν σε αυτό το σύμφωνο επανεγκατάστασης. Γι' αυτό λυπούμε και θέλω να το πω. Την, ε, λυπούμε για την αποχώρηση των ΙΠΑ από το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Μια μεγάλη χώρα η οποία έχει μια μακρά παράδοση επανεγκατάστασης και η οποία θα μπορούσε να έχει αποτελέσει θετικό παράδειγμα για άλλες χώρες. Επίσης, καλωσορίζω όλα τα επιχειρησιακά μέτρα που έχουν προταθεί όσον αφορά την υποδοχή και την εισδοχή. Μια πιο συντονισμένη προσέγγιση είναι πολύτιμη για την ασφάλεια όλων μας. Σωστή έλεγχη των αφήξεων και χρήση των βάσεων δεδομένων είναι σημαντικά στοιχεία για να διαχειριστούμε καλύτερα τις ροές και να αξιολογήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό έχει σημασία κλειδί για να ταυτοποιήσουμε τους ευάλωτους ε, πρόσφυγες, ειδικά τα παιδιά, και να έχουμε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Η ουσία του συμφώνου είναι ότι δεν μπορούμε να ευσυχάζουμε ε, όσον αφορά το μέλλον. Ναι, συλλογικά έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες για να στηρίξουμε και τους πρόσφυγες αλλά και τις γειτονικές χώρες ε, που επηρεάζονται από την σύγκρουση στην Σύρια. Αλλά η σύγκρουση αυτή δεν έχει τελειώσει. Δυστυχώς. Και καταστάσεις όπως η κρίση των Ροχίνγκια μας υπενθυμίζουν πως έχουμε άλλες κρίσεις ε, παραλλήλου που θα εμφανιστούν ανά τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και έρχομαι τώρα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Ενώ πρόσφατα εστιάζουμε στους πρόσφυγες, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που μετακινούνται σήμερα δεν είναι πρόσφυγες. Η κινητικότητα θα καθορίσει το μέλλον και τους καιρούς μας. Έχει ακουστεί ότι η εποχή μας ε, θα ονομαστεί από του ιστορικού του μέλλοντο ω η εποχή της ανθρώπινης κινητικότητα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα την σταματήσουμε, αλλά πώς θα την διαχειριστούμε καλύτερα από κοινού. Πριν από δύο ώρες ε, συναντήθηκα με τους δύο διαμεσολαβητέ ε, που έχουν στόχο την σύνταξη του Παγκόσμιου Συμφώνου για ασφαλιόμαλη και έφτακτη μετανάστευση και εξέφρασα τις ευχαριστίες μου για το αρχικό σχέδιο κειμένου, το οποίο αποτελεί μια καλή βάση διαπραγματεύσεων. Και εξέφρασα την άποψή μου ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο θα είναι αποτελεσματικό, αν διακρίνει σαφώς μεταξύ έφτακτης και παράτυπης μετανάστευσης. Για να κάνουμε λοιπόν ένα βήμα προς τα εμπρός, Όλες οι χώρες οφείλουν να αναγνωρίσουν ε, στο πλαίσιο αυτού του Παγκοσμίου Συμφώνου πως πρώτον οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να υποδεχτούν κάποιους ανθρώπους στην επικρατειά τους. Δεύτερον, οι χώρες προέλευσης ε, θα πρέπει να ε, δεχτούν τους δικούς τους υπηκόους οι οποίοι έχουν μετακινηθεί παρατύπως. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την δημογραφία αλλά ούτε και την οικονομία. Η διευκόλυνση της νόμιμης οικονομικής μετανάστευσης είναι ένα μέσο, μεταξύ άλλων, για να διαχειριστούμε καλύτερα τη μετανάστευση. Εάν την διαχειριστούμε σωστά, αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, για τους εν λόγω μετανάστες και για τις χώρες προέλευσης. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με κράτη-μέλη για να αναπτύξουμε στοχευμένα πιλωτικά έργα νόμιμης μετανάστευσης με συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, η οικονομική κατάσταση στις χώρες υποδοχής ε, και η, και η ικανότητα ένταξη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπως και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης. Επίσης έχουμε υποχρέωση να λάβουμε στα σοβαρά την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει αξιοπρεπής δουλειά για τους μετανάστες οι οποίοι κατοικούν νομίμως στην επικράτεια. Πρέπει επίση να είμαστε ειλικρινεί. ρεαλιστέ. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν πρέπει να επιστραφούν το των δυνατόν οι πολίτες μας. Θέλουν αποτελέσματα σε αυτό το μέτωπο. Μπορούμε να έχουμε και να επιδείξουμε φιλοξενία σε αυτούς οι οποίοι τη χρειάζονται, μόνο εάν η φιλοξενία αυτή δεν γίνεται αντικείμενο κατάχρησης από αυτούς που δεν τη χρειάζονται το Παγκόσμιο αυτό σύμφωνο θα πρέπει να δει και τις αιτίε της παράτυπης μετανάστευσης και στο πλαίσιο αυτό έχει μεγάλη σημασία η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει ξεκάθαρα να διατυπώνει μια υποχρέωση για τις χώρες προέλευσης να δέχονται τους υπηκόους τους πίσω. Η Ευρώπη ήδη είναι σε επαφή με τρίτες χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Γουινέα και η Αιθιοπία για να συζητήσει ζητήματα επιστροφών και επανεισδοχής. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση θα πρέπει να στηρίξει και να ενισχύσει περαιτέρω την πρόοδο αυτή. Τέλος, πρέπει να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να μείνουν στις χώρες μας, είτε είναι πρόσφυγες, είτε άλλοι νομίμως διαμένοντες μετανάστες, πρέπει να βρουν την θέση τους και τον ρόλο τους στις κοινωνίες μας. Η επένδυση στην ένταξη είναι και προς το κοινωνικό και το οικονομικό μας συμφέρον, αν θέλουμε να έχουμε συνεκτικές κοινωνίες για το μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και τα δύο αυτά σύμφωνα έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Κλοντ που διοργάνωσε την σημερινή συνεδρίαση. Είναι πραγματικά μια ιστορική συνεδρίαση. Πρέπει να είμαστε τολμηροί και φιλόδοξοι για το μέλλον, πολιτικά, επιχειρησιακά και οικονομικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να μιλήσουν με μία φωνή στην διεθνή αρένα, στην διεθνή σκηνή για να επιτύχουμε ένα φιλόδοξο παγκόσμιο σύμφωνο μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κοινή παγκόσμια συνεννόηση για τη διαχείριση των ροών προσφύγων και μεταναστών παγκοσμίω. Επίσης βασίζομαι σε εσάς ε, για να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις σας για τα δύο σύμφωνα αυτά. Εγώ βεβαίω θα ενημερώνω πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως κάνω πάντα και ευχαρίστως ε, θα έρθω να ξανασυζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς ε, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, όπως υπογραμμίσατε και εσείς ε, με απόλυτη συνοχή. Αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολα είναι και τα δύο σύμφωνα και στην εφαρμογή τους. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την κεντρική ομιλία και περνάμε στο πρώτο κομμάτι της συνόδου, στην πρώτη συνεδρία, πριν περάσουμε στη συζήτηση με τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Περνάμε στο πρώτο κομμάτι της διαδικασίας. Έχουμε εκπροσώπους από τα Ηνωμένα Έθνη, από τις με κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, οπότε σας παρακαλώ να έρθετε εδώ. Και θα ήθελα ξανά για μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Επιτροπό. Uh, και έχουμε εκπροσώπους επίσης και από την Αγία Έδρα. Περιμένουμε μέχρι να ανέβουν στο βήμα. So, colleagues, as, um, so as not to, uh... Αγαπητοί συνάδελφοι, για να μείνει χρόνος και για τη συζήτηση με εσάς, ε, θα κάνω εγώ μια εισαγωγή καθώς ε, έρχονται οι συνάδελφοι στο βήμα. Okay, so welcome to all of you and uh, this first session which will... Καλώς ορίσατε σε αυτό το πρώτο κομμάτι της Συνόδου και μετά από αυτό θα κάνουμε τη συζήτηση με τους εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί με τους συνεισηγητές μας, την κυρία Κιέγγι και την κυρία Μέτσολα, που είναι εισηγήτριε για την ολιστική μας προσέγγιση για τη μετανάστευση. Πριν από αυτή τη σημαντική συζήτηση, ε, με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τους ειδικούς μας προσκεκλημένους ε, που θα μας παρουσιάσουν τις δικές τους ε, απόψεις, τη δική τους εικόνα ε, για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα και για την πρόοδο που θεωρούν ότι έχει σημειωθεί και χαίρομαι που συνεργάζονται μαζί μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί μας. Ε, ε, να καλωσορίσω λοιπόν τον Βόλκερ Τέρκ, βοηθό είπα του αρμοστή για την προστασία του UNHCR, τον Λιονόρ Νιέτο Λιόν, ε, την ε, κυρία Λεωνόρ Νιατολιών, επικεφαλής μονάδα ΕΚΟ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Σπασία Παδοπούλου, ανώτερη υπευθύνη πολιτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις πρόσφυγες και του Εξόριστου, και ο πατήρ Φάμπιο Μπάτζο, υπογραμματέας ε, του Τμήματο Μεταναστών και Προσφύγων τη Αγία Έδρα. Σα καλωσορίζω όλου. θερμά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μα παρουσιάσετε και τι δικέ σα απόψει. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως υπενθύμηση η διακήρυξη της Νέας Υόρκης αφορά κάποιες πρακτικές ε, πτυχές ε, και ένα σχέδιο μηδέν. Και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο πρεσβείς που τους ανέφερε και τους δύο επίτροπους ε, που θα μιλήσουν στην επόμενη συνεδρία. Αυτό το σχέδιο μηδέν θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις και τις επίσημες συνομιλίες και αποτελείται από δύο κομμάτια. Όλοι μας οι ομιλητές θα μιλήσουν και για τα δύο αυτά σχέδια και θα ακολουθήσει συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θα ζητήσω από τον κύριο Βόλκερ Τούρκ, ε, βοηθό υποτορμοστή από την UNHCR, να μας παρουσιάσει τη δική του, ε, την προσέγγιση της ΥΠΑ ε, στο για τους πρόσφυγες της UNHCR. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ με αυτή την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας, ε, μέσα στου βουλευτέ, για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και το οποίο, για να το δούμε με απόλυτη ε, με απόλυτο ρεαλισμό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο και εμείς ε, υπολογίζουμε στην υποστήριξη όλων και ειδικότερα στην υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι και σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο η Διακοινοβουλευτική Ένωση έχει συνεργαστεί πολύ για τα ζητήματα της μετανάστευσης και το προσφυγικό. Θα ήθελα να εστιαστώ φυσικά στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Μετανάστες και πριν μπω σε κάποιες από τις λεπτομέρειες θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω το γενικό πλαίσιο ε, μέρος του οποίου ήδη μας περιέγραψε ο Επίτροπος κ. Σαβραμόπουλος, αλλά ήθελα να σας το παρουσιάσω και εγώ από την πλευρά ε, του Οργανισμού των Ηνωμένων για τους ε, πρόσφυγες και είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε αυτή την εικόνα του παγκόσμιου πλαισίου. Έχει παρατηρηθεί μεγέθυνση του μεγέθους της πολυπλοκότητας του εύρους ε, ε, του φαινομένου αυτού τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό μας το δείχνουν τα νούμερα. αλλά καθίσταται σαφές και από την εκτεταμένη φύση του εκτοπισμού. Όταν μιλάμε για 22,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Μιλάμε για ανθρώπους που ξεφεύγουν από συγκρούσεις, σειράξεις, βία, διώξεις, ε, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλο και περισσότερο παρατηρούμε να συνδυάζεται αυτό με ζητήματα όπως υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή. Παρότι αυτά μπορεί να μην είναι η βασική αιτία, ε, αφορμή για τον εκτοπισμό, παίζουν σημαντικό ρόλο σε χώρες όπως ε, η Σομαλία, η Αιθιοπία, χώρες στο κέρας Αφρικής αλλά και σε άλλα μέρη. Και είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Επίσης είναι σημαντικό ειδικότερα ε, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνομιλιών να θυμόμαστε ότι οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από όλα αυτά τα φαινόμενα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη, αλλά στο Νότο. 84% αυτών βρίσκονται στα πιο ε, φτωχά μέρη του κόσμου και έχουν να αντιμετωπίσουν ε, αναπτυξιακά προβλήματα, ιδιαίτερα σε χώρες όπως ε, στην Ουγγάντα, από όπου έχει φύγει ένα τους τελευταίους μήνες, όπου έχει μπει ένα εκατομμύριο ε, τους τελευταίους μήνες πολίτες από τον Νότιο Σουδάν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις υποδομές, για τις κοινότητες, για την ένταση της ανθρωπιστικής πίεσης και των απαιτήσεων. Ένα άλλο στατιστικό στοιχείο σημαντικό είναι ότι το 60% όλων των προσφύγων είναι στην πραγματικότητα φιλοξενούμενοι σε 10 χώρες όλες και όλες. Κάτι που μας δείχνει πόσο μεγάλη έλλειψη ισορροπίας παρουσιάζει το παγκόσμιο σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε. Ξέρουμε επίσης το θέμα δεν είναι μόνο θέμα προσφύγων αλλά και θέμα ανθρώπων εσωτερικά εκτοπισμένων. Περίπου ε, αρκετά εκατομμύρια και περίπου 10, 10 εκατομμύρια πάτριδες και όπως ακούσαμε και από τον Επίτροπο κύριε Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο της Μιανμάρ και του Μπαγκλαντές, ε, το ότι έχουμε πάνω από 700.000 πρόσφυγες ε, Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ που έχουν διαφύγει στο Μπαγκλαντές και αυτό είναι αποτέλεσμα του καθεστώτος ε, του απάτριδος για αυτούς τους ανθρώπους και της σοβαρής διακριτικής μεταχείρισης πέραν όλων των υπόλοιπων παραβιάσεων. Λόγω όλων αυτών το 1946 ένα από τα πρώτα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης κατέστησε σαφές ότι οι πρόσφυγες είναι διεθνές ζήτημα, επηρεάζουν στο σύνολό της τη διεθνή κοινότητα, έχουν διεθνή χαρακτήρα και απαιτούν διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίζετε το σχετικό, να αντιμετωπίζετε τα σχετικά προβλήματα. Αυτή η αναγνώριση εντός των ΗΕ έγινε πολύ νωρίς και αναγνωρίστηκε σαφέστατα η ανάγκη να γίνει κάτι γι' αυτό. Από το 46 λοιπόν και μετά παρατηρούμε ότι στα θέματα το προσφυγικά στη διεθνή αρένα υπάρχουν σαφείς, σαφή πολιτικά και επιχειρησιακά πλαίσια που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των προσφύγων. Το παρατηρούμε αυτό όχι μόνο σε νομικό και θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στη δημιουργία θεσμών, όπως το UNHCR, ε, και όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη. Και το τελευταίο που βλέπουμε είναι η διακήρυξη της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρατε. Είναι σημαντική η διακήρυξη της Νέας Υόρκης, διότι γέννησε δύο διαδικασίες, όπως αναφέρατε, δύο προϊόντα. Το ένα αφορά τους πρόσφυγες και το άλλο την ασφαλή ομαλή και εύθεκτη μετανάστευση. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, ε, το UNHCR εκεί λειτουργήσε υβριδικά ουσιαστικά. Η πατιαρμοστία ζήτησε φέτος ε, βάση της πρακτικής εφαρμογής ε, του συνολικού πλαισίου, του πλαισίου ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού σε πολλές χώρες στον κόσμο και βάση της εμπειρίας που είχαμε και μετά από διαβούλευση με όλους ενδιαφερομένους, κράτη-μέλη, βουλευτές, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τοπικές κοινότητες, ώστε να προκύψει κάποιο κείμενο και τώρα βρισκόμαστε προς το τελευταίο κομμάτι αυτής της διαδικασίας έχοντας ε, αντλήσει διδάγματα από τις 13 ε, χώρες όπου έχει εφαρμοστεί το CRF. Έχουν γίνει διάφορες διαβουλεύσεις πέρυσι στη Γενέβη. Επίσης είχαμε και πολλές περιφερειακές διαβουλεύσεις φυσικά. Και ξεκινήσαμε να εκπονούμε το σχέδιο 0 του Παγκοσμίου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες που εκδόθηκε στις 31 Ιανουαρίου και ξεκινήσαμε τις επίσημες διαβουλεύσεις ε, γύρω από εκείνη την ημερομηνία στη Γενέβη με κράτη-μέλη και με άλλους ενδιαφερομένους ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες θα εμπλουτιστεί και θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις χώρες που επηρεάστηκαν από αυτά τα φαινόμενα, αλλά και ότι θα χαρακτηρίζεται από αυτή την κοινή βούλευση που εξέφρασε ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος, αλλά και που πολλές φορές έχετε εκφράσει πολλά μέλη εδώ της Επιτροπής σας, ε, αυτή την ανάγκη να προχωρήσουμε. Τι σημαίνει αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο, το σχέδιο 0. Να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Κατ' ουσίαν προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα αιώνια κενά που αντιμετωπίζουμε την, ε, το διεθνή επιμερισμό των ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Αναφέρεται στο προήμιο της, ε, του Συμφώνου του 1951, αλλά πουθενά δεν διατυπώνεται λεπτομερώς. Απλά αναφέρεται η ανάγκη διεθνού συνεργασία. Αλλά το πώ θα επιτευχθεί, πώ θα εφαρμοστεί, ποιο θα έχει την ευθύνη για όλο αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Ε, σε αρκετές λεπτο... αρκετά αναλυτικά. Αλλά εδώ αντλούμε από χρόνια εμπειρία ουσιαστικά, πάνω από 50 και το Παγκόσμιο Σύμφωνο ουσιαστικά προσπαθεί να θεσπίσει τα μέτρα υποστήριξης που χρειάζονται οι χώρες οι οποίε έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση λόγω τη τεράστια ροή, όπως η Ουγγάντα, η Τανζανία, η Αιθιοπία και άλλες ή λόγω μιας παρατεταμένης κατάστασης ε, ε, στην οποία βρισκόνται για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αφορά ειδικότερα τους 5,3 εκατομμύρια Σύρους ε, πρόσφυγες στις διάφορες χώρες. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να εμπλακούν ε, περισσότερες χώρες, όχι απλά οι χώρες πάνω στις οποίες βασίζεται η διεθνής κοινότητα, ε, που είναι συχνά οι χώρες χορηγοί όπου διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αφορά και θέματα όπως η επανακατάσταση. Η επανακατάσταση είναι ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης το οποίο είναι αναγκαίο. Αναγκαίο όχι μόνο για καταστάσεις που βρίσκονται γύρω από την Ευρώπη αλλά και στο πλαίσιο ε, χρήσης του ως ενός καθολικού εργαλείου ε, επιμερισμού αλληλεγγύης. Με την Παγκοσμία Τράπεζα από την άλλη έχουμε αντλήσει μεγάλη εμπειρία από την αναπτυξιακή, μέσω της αναπτυκής βοηθείας. Γνωρίζουμε από εμπειρία μας ότι όταν οι πρόσφυγες παραμένουν στην ίδια κατάσταση για πολύ καιρό θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ε, έγκαιρη άφηξη, ε, έλευση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας ώστε να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, σε υπηρεσίες που να παρέχονται όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για τις κοινωνίες υποδοχής ώστε κάποιες από τις αναγκαστικές εκτοπίσεις, κάποιους από τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς να μετατρέπονται σε αναπτυξιακές προοπτικές. Εκεί λοιπόν εστιαζόμαστε περισσότερο στην αναζήτηση λύσεων διότι όπως ξέρετε έχουν λείψει ε, λύσεις πολλές φορές, εδώ και καιρό, ειδικότερα όσον αφορά τον εθελοντικό επαναπατρισμό. Αλλά ελπίζουμε ότι εστιάζοντας την αντιμετώπιση των ε, ριζικών αιτιών ε, και όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας εστιαζόμενοι στην πρόληψη, στην εξέβρεση πιο δημιουργικών τρόπων αντιμετώπισης των αιτιών ελπίζουμε ότι έτσι θα στηρίξουμε ισχυρότερα εκ μέρους της διεθνής κοινότητας όλα αυτά τα ζητήματα. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Μετανάστες ε, είναι νομικά μη δεσμευτικό. Δεν είναι νέα συνθήκη ούτε σύμβαση. Ωστόσο ταυτόχρονα θα έχει ύψιστη πολιτική σημασία γιατί θα υιοθετηθεί και από τα 193 κράτη-μέλη. Και εφόσον υιοθετηθεί ε, προφανώς θα αποτελέσει το άλμα αλλαγή που χρειαζόμαστε, διότι ολόκληρη η διεθνή κοινότητα θα βοηθήσει τι χώρε που ε, χρειάζονται βοήθεια. Αυτό με φέρνει πίσω σε αυτά που επιχειρείτε κι εσείς ε, στο λειτουργήμά σας ως βουλευτές. Ε, για μας αυτό που θα ήταν πολύ σημαντικό θα ήταν να εκφράσουμε ισχυρή υποστήριξη. Να εξασφαλίσουμε να, την αναγνώριση του παγκόσμιου χαρακτήρα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ζητήματος. Να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι δεν βρίσκεται εκτό όλων αυτών, αλλά ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Το βλέπουμε αυτό και εκ μέρου των κρατών μελών, αλλά και εκ μέρου των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τη Κομισιόν. Θέλουμε επίση να εξασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση μέσων, εργαλείων. Ξέρω ότι και εσεί ω Ευρωβουλευτέ ε, φυσικά ε, έχετε τον έλεγχο του προπολογισμού όσον αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, για παράδειγμα, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό που ξεκίνησε στο πλαίσιο τη δημοσιονομική διαδικασία από τον Επίτροπο είναι να ληφθεί υπόψη αυτή η διάσταση ε, του εκτοπισμού και ότι και αυτό, για αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να στείλουμε ένα ε, ηχηρό μήνυμα διότι να ακούσουμε τα μηνύματα που ακούμε από τις διάφορες χώρες ε, υποδοχή ακούμε ότι ναι καλά είναι όλα αυτά τα, κύμα, τα κείμενα αλλά χρειάζονται περισσότερη δέσμευση από άλλα μέρη του κόσμου να υπάρξει επιμερισμός των ευθυνών στο πλαίσιο του προσφυγικού και του μεταναστευτικού και τι μπορείτε να κάνετε για να γίνουν τα πράγματα πιο προβλέψιμα στον τομέα της χρηματοδότηση, στον τομέα τη αναπτυξιακής βοήθεια, λαμβάνοντα υπόψη αυτό τον εκτοπισμό. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της επανεγκατάστασης, ε, καθώς επίσης και των συμπληρωματικών διάβλων, εναλλακτικών διάβλων ε, ε, υποδοχής. Βεβαίως, όσον αφορά τα θέματα αυτά, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα ακόμα. Χρειαζόμαστε αντιμετώπιση με αυτόν τον τρόπο και στην Αφρική και στην Σύρια. Για τις πιο ευάλωτες περιοχές θα πρέπει να βρούμε τρόπους πρόσβασης ασφαλούς πρόσβασης σε γειτονικές ε, χώρες. Ε, μιλάμε εδώ για πολλές χιλιάδες ανθρώπους που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν. Για την ώρα είναι πολύ χαμηλή αριθμή, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. Ε, τελευταίο ζήτημα, το συζητάτε και εσείς, το κοινό σύστημα ασύλου, το συζητάτε στην Επιτροπή Ελευθεριών του Κοινοβουλίου. Ε, λέμε λοιπόν ότι οτιδήποτε αποδεικνύει την εξωτερική αλληλεγγύη, ε, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ε, κάποιοι μηχανισμοί αλληλεγγύης που συζητάτε, συμπεριλαμβανομένου και των συστημάτων επανεισδοχής. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο. Και μεταβδίδουν το μήνυμα ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλύπτει το άσυλο, προστατεύει το άσυλο με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ε, προωθείται ως αξία η οποία θα πρέπει, την οποία δεν θα πρέπει να λησμονούμε. Οι διαβουλεύσεις ε, με τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει, θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Ευελπιστούμε ότι θα έχει η διαδικασία μέχρι τον Ιούλιο και ευελπιστούμε ότι το κυρίαρχο ζήτημα της ε, ε, εξέβρεσης ισορροπίας από τη μία πλευρά του εθελοντικού χαρακτήρα του κειμένου και από την άλλη πλευρά ε, η ανάγκη δέσμευσης ε, θα βοηθήσει έτσι ώστε ε, οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα θα βοηθηθούν ιδιαίτερος και μπορώ να σας πω ότι αυτή η εξέβρεση ισορροπίας θα είναι ακριβώς για τους επόμενους μήνες το πιο δύσκολο, το πιο δυσχερές στοιχείο. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την έννοια των λεγόμενων μου ε, έχει παίξει, παίζει και θα εξακολουθήσει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά ήθελα να πω και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Μας μεταφέρατε την σκοπιά του ΟΗΕ. Μία επενθύμηση για τους εθνικούς ε, βουλευτές. Ε, αν δεν έχετε συμπληρώσει το χαρτάκι και θέλετε να πάρετε το λόγο, συμπληρώστε το έντυπο. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει τον λόγο και είμαι φυλακτικό γιατί πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή και η πρώτη συνεδρία. Λοιπόν, μπορείτε σε 8 λεπτά να πείτε αυτά που θα λέγατε σε 15 και μετά τα 8 λεπτά δεν ακούει και κανείς ούτως ή άλλως. Οπότε περιοριστείτε σε 8 λεπτά σας παρακαλώ γιατί έχουμε πολύ κόσμο που θέλει να μιλήσει. Εάν δεν έχετε ακόμα συμπληρώσει το χαρτάκι, συμπληρώστε το, δώστε το στον κλητήρα και θα κλείσω σε 5 λεπτά τον κατάλογο των ομιλητών. Κατόπιν λοιπόν έχουμε την ε, κυρία Λιόν ε, από... Α, εσείς είστε. Α, συγγνώμη, δεν είχαμε συναντηθεί από την Κομισιόν. Αυτά που είπα για τα 8 λεπτά ισχύουν και για σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ε, εθνικοί βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέρος ε, στη συγκεκριμένη συνεδρία. Θα ήθελα ε, να ξεκινήσω επενώντας την πρωτοβουλία αυτή, τα είπε και ο Επίτροπος ο κύριος Αβραμόπλος, αλλά θεωρώ ότι η πρωτοβουλία της σημερινής συνάντησης σήμερα είναι πολύ επίκαιρη αμέσως ε, μετά την δημοσίευση των δύο σχεδίων συμφώνων και πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Θα ήθελα να επενέσω και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, όπως ανέφερε εδώ πέρα και ο βοηθός ύπατος ε, αρμοστής ε, του ΟΗΕ για το ότι υπάρχει μια σταθερή προσήλωση στις αρχές που αναφέρουν τα σύμφωνα αυτά. Η έγκριση της δήλωσης της Νέας Υόρκης για πρόσφυγες και μετανάστες ε, το 2016 ήταν ε, ένα ορόσημο για το θέμα της μετανάστευσης και του εκτοπισμού. Μέσω της δήλωσης αυτής η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε για την βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης και για τον καλύτερο διαμοιρασμό της ευθύνη. Οι αριθμοί των προσφύγων και των ετούντων άσυλο είναι συγκλονιστικοί τα ανέφερε και ο εκπρόσωπος ε, του ΟΗΕ και πιθανώς ε, θα αυξηθούν ε, ως αποτέλεσμα νέων συγκρούσεων και των παλαιών επίσης. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τις Πρόσφυγες λοιπόν παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα της αντίδρασης στην κατάσταση αυτή. Για πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα εταιρό κλειδί τη υπατσαρμοστίας του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση τη κατάσταση των προσφύγων εδώ και χρόνια. Σημαντικό κομμάτι του προπολογισμού ανθρωπιστική βοήθεια τη Κομισιόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαινε ακριβώ σε τέτοια ζητήματα σε πολλέ χώρε. Στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ουγγάντα, στην Κένια, το Ιράκ. Έχουμε παρέμβει σε αυτές τις καταστάσεις για να δώσω μόνο λίγα παραδείγματα και θα ήθελα με τη να επενέσω και τις ε, τρομερές προσπάθειες που έχουν κάνει οι χώρες οι οποίες φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Ε, επιπροσθέτως ε, προς την χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει και νέες πολιτικές στον τομέα αυτόν. Τον Απρίλιο του 2016 η Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση για τον εκτοπισμό και την ανάπτυξη. Στα πλαίσια της παγκόσμιας ανθρωπιστικής διάσκεψης που έγινε τον Μάιο του 2016 στην Κωνσταντινούπολη. Η πολιτική αυτή είχε ως αφετηρία την εμπειρία ετών και σε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και σε πρόσφυγες. Η προσέγγιση η οποία απλά επέτρεπε στους πρόσφυγες να επιβιώσουν πλέον δεν μπορούσε να διατηρηθεί δεδομένη της διάρκειας της μέσης κρίσης ε, την σήμερον ημέρα. Γι' αυτό προτείναμε μία ε, πρόταση η οποία είχε ως στόχο να μην παραταθεί ο εκτοπισμός ε, και αφορά και την ανάπτυξη ανθρωπιστικής δράσης και πολιτικών φορέων για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του εκτοπισμού και να ανταποκριθούμε και στις ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων που φιλοξενούν. Κουνθεί μια προσέγγιση η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών που θα συνεισφέρουν στις ε, κοινότητες που τους φιλοξενούν μέχρι να βρεθούν οι προϋποθέσεις μιας μόνιμης λύσης. Αντιμετωπίζουμε τώρα και αναπτύσσουμε αυτή την στρατηγική επιτόπου στα διάφορα πεδία. Και βεβαίως έχουμε και την το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προσφύγων και το προσχέδιο Παγκόσμιου Συμφώνου. Προσπαθώ τώρα να μην επαναλάβω όλα όσα είπε ο κύριος Επίτροπος. Θα ήθελα να κάνω κάποιες συγκεκριμένες γενικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της ε, του ΟΗΕ στο πλαίσιο αυτό και στην ανάπτυξη του συμφώνου και δράτωμα της ευκαιρίας ε, να επενέσω και τον ρόλο της υπατσαμουστίας μέχρι στιγμή στην διαδικασία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει και την δέσμευσή της ε, για, στο, στην σύμβαση για το καθεστώς ε, των προσφύγων και το σχετικό πρωτόκολλο ως τη βάση αντιμετώπισης ε, του ζητήματος των προσφύγων. Επίσης έχουμε και το σχέδιο δράσης ε, και την συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των προσφύγων, όπως ήδη ανέφερε ο Επίτροπος. Σε σχέση με το σχέδιο πρόγραμματος ε, δράσης, εκτιμούμε το ότι είναι ακριβώς ένα επιχειρησιακό πλαίσιο αντιμετώπισης του ζητήματος. Η αντιμετώπιση λοιπόν των αιτίων του εκτοπισμού ε, συνολικές μακροπρόθεσμες απαντήσει. Ε, Διαμερισμό τη ευθύνη. Ε, διεθνή συνεργασία, αλληλεγγύη, η εμπλοκή των διαφόρων μερών και μόνιμες και διαρκεί λύσεις είναι βασικά στοιχεία που αναφέρονται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο περί προσφύγων. Στους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπλακεί επικοδομητικά στις διαβουλεύσεις που θα λάβουν χώρα και ελπίζουμε πραγματικά η διαδικασία αυτή να οδηγήσει σε μια επιτυχή έγκριση του Παγκόσμιου Συμφώνου, ε, ένα μέσο το οποίο, όπως τόνισε και ο κύριος Αβραμόπουλος, πλέον απαιτείται περισσότερο από ποτέ. Νομίζω ότι περιορίστηκα και σε λιγότερο χρόνο. Σε 7-8 λεπτά καταφέρατε να πείτε αυτό που θα λέγατε σε 12. Βλέπω ότι τηρείται ε, τους χρόνους που ζητήσαμε και έτσι θα μας μείνει και χρόνος ε, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να κάνει ερωτήσεις ε, και εγώ δεν θα λέω πω συμπεράσματα, σας το υπόσχομαι. Ακολουθεί η κυρία Παπαδοπούλου από την ΕΚΡΑ. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με προσκάλεσετε σε αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση σήμερα. Θα σας δώσω την άποψη των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη συζήτηση και θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που ήδη κυκλοφορούν στην κοινότητα των ΜΚΟ και στις επίσημες διαβουλεύσεις στη Γενέβη. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αναγνωρίζουμε τις τεράστιες προσπάθειες του UNHCR και την πρόοδο προς το Παγκοσμίο Σύμφωνο. Εκτιμάμε ιδιαίτερα τη διαρκή χωρίς αποκλεισμούς δέσμευση των ΜΚΟ και τη συμμετοχή του στο τελευταίο έτος. επίση. αναγνωρίζουμε τη διαρκή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ε, διακήρυξης τη Νέα Υόρκης, τη συνομιλίες ε, και σε θέματα όπω η αναγκαστική, ο σεκτοπισμός όπως αναφέραμε και για την ε, ενίσχυση της υποστήριξης. Καλωσορίζουμε το σχέδιο 01 τη προγραμματική δράση και πιστεύουμε ότι καλύπτει τα πάντα, σχεδόν όλα τα σημαντικά ζητήματα πολλά θετικά στοιχεία περιλαμβάνει, τα οποία επικροτούμε, τα οποία δείχνουν ότι σταδιακά αλλάζει η προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας. Απομακρυνόμαστε από τις ε, κατασκηνώσεις ε, και τη διαρκή συντήρηση σε ένταξη στις τοπικές κοινότητες, σε αυτονομία, ανεξαρτησία των προσφύγων. Αυτό είναι μια αλλαγή μοντέλου αντιμετώπισης θα έλεγα. Η αναγνώριση ότι είναι απαραίτητο οι πρόσφυγες να εργαστούν και ότι αυτό αποτελεί δικαίωμά τους είναι πλέον μια πιο παγιωμένη αρχή στο πρόγραμμα δράσης όπω επίση και η ενίσχυση των σχέσεων με αναπτυξιακού παράγοντε όπω η Παγκοσμία Τράπεζα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, πολύ θετικά στοιχεία που μα κάνουν να ελπίζουμε πολλά. Ταυτόχρονα, αν θέλουμε το Παγκοσμίο Σύμφωνο όμω να μεταμορφώσει την προσέγγιση της διεθνού κοινότητα όσον αφορά την προστασία, πράγμα το οποίο ελπίζουμε, χρειάζονται ακόμα δύο πράγματα, τα οποία εμείς θα θέλαμε να επισημάνουμε. Πρώτον, η ανάγκη ανάπτυξης ε, μιας συλλογική φιλοδοξίας ε, εντό του σχετικού πλαισίου και με στόχους συγκεκριμένου και δεύτερον χρειάζεται να γίνουμε λίγο πιο επιχειρηματικοί, να παρέχουμε καθοδήγηση στα κράτη για το πώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεράστιες ροές και να βοηθήσουμε να παρασκευθούν λύσεις προς τους πρόσφυγες ε, παγκοσμίω. Αυτά θα αναλύσουμε για τη συλλογική φιλοδοξία. Πάμε πίσω για λίγο στους στόχους του Παγκοσμίων Συμφώνων που ήδη ανέφερε ο Φόρκερ Τέρκ. Στο πλαίσιο του UNHCR θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό που υπήρχε ανέκαθεν όπως αναφέρθηκε στο Διεθνή Σύστημα Προστασίας των Προσφύγων ε, ώστε να διασφαλιστεί ε, προβλέψιμος ε, επιμερισμός παγκόσμιας ευθύνης. Αυτός ο επιμερισμός της ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι που θα προσθέσει αξία σε όλα αυτά ιδανικά θέλουμε ένα καλύτερο ορισμό. Τι εννοούμε ε, παγκόσμιος επιμερισμός της ευθύνη. Περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτό θέλουμε. Πώς μεταφράζεται δηλαδή στην πρακτική. Στην υποδοχή, στην εισδοχή, στην κάλυψη αναγκών των κοινοτήτων υποστήριξης, ε, με την παροχή λύσεων, δεσμεύσεων για την επαναγκατάσταση. Αλλά υπάρχουν αλλά συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να εμπλέκονται περισσότερα τα κράτη, περισσότερα κράτη πρέπει να υπάρχουν περισσότερη, μεγαλύτερη βούληση ε, και υποχρεώσεις παρά απλά υποσχέσεις. Και ο Φόλκερ ήδη έχει ακολουθήσει, έχει, έχει λάβει τέτοια σχόλια από τη ΜΚΟ και γνωρίζει όλες αυτές τις απαιτήσει. Το δεύτερο όμως που απαιτείται είναι να έχουμε και ένα ε, παγκόσμιο εύρος, ε, διότι τώρα μιλάμε ότι οι σημαντικοί φορείς είναι τα κράτη και δεν βλέπουμε να υπάρχει συλλογική ευθύνη, δηλαδή να υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι πρόσφυγες του κόσμου φιλοξενούνται στον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά, στον πρώτο κόσμο, αλλά και η Ευρώπη, ε, τα κράτη του πρώτου κόσμου είναι χώρες υποδοχής, δεν είναι μόνο χορηγοί. Οπότε θέλουμε συλλογική ευθύνη να αναπτυχθεί μέσω του προγράμματος δράσης το τρίτο που απαιτείται, είναι να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά το δικαίωμα ασύλου και μη επαναπρόθεσης. Το πρόγραμμα δράση θα μπορούσε να παρέχει ισχυρότερη υποστήριξη και προστασία όσον αφορά τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ε, διασφάλιση του δικαιώματο αίτηση ασύλου, πρόσβαση στα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά ήδη στο προήμιο, εκύρωση της ε, σύμβαση τη Γενέβη από όλα τα κράτη-μέλη Αυτά ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα ώστε να συμπεριληφθούν όλα αυτά στο κείμενο θα θέλαμε. Αυτά όσον αφορά τη συλλογική φιλοδοξία. Για τη δεύτερη πτυχή, την πιο έντονη ε, δράση. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε κάπως υβρεδικά, συνδυάζουμε αρχές με κάποια καθοδήγηση σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στην αναθεώρηση λοιπόν που ήδη έχει ξεκινήσει, καλό θα ήταν ορισμένα από αυτά να αποτελέσουν καθοδήγηση, να μεταφραστούν σε καθοδήγηση προ τα κράτη-μέλη, ώστε να γνωρίζουν τι να κάνουν σε επιχειρήσει μεγάλη κλίμακα, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τον επιμερισμό των ευθυνών, για τι σχετικέ διευθετήσει, ξεκινώντα από το βραχυπρόθεσμο μέχρι το μακροπρόθεσμο, ε, προγραμματισμό για περιπτώσει έκτακτη ανάγκη, οργάνωση υποδοχή, με συγκεκριμένη ε, καθοδήγηση, ε, την όλη κοινωνική προσέγγιση που θα έπρεπε να που χαρακτηρίζει όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει και που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά θα μπορούσαν να δομηθούν καλύτερα ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιούν όλα αυτά τα πράγματα καλά. Τι σημαίνει ουσιαστικά προσέγγιση όλης της κοινωνίας, πώς συντονίζεται, πώς ε, ε, θα έχει κανείς και τη συμμετοχή ε, συστηματικά των προσφύγων. Ουσιαστικά πώς οι εθνικές διευθετήσεις με σαφή ε, κίνητρα, με σαφείς στόχους, με σαφή ηγεσία, πώς θα υλοποιούνται. Επίσης αξιόπιστα συστήματα παρακολουθήσεις και αξιολόγησης που ήδη προβλέπονται φυσικά στο πρόγραμμα δράσης, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί εμείς ε, αργότερα στο έτος ε, και να παρουσιάσουμε συγκεκριμένους στόχους, περιθώρια χρονικά θα μπορούσαμε να τα συνδέσουμε στους ε, ε, αναπτυξιακούς στους στόχους ανάπτυξης, βιώσιμης ανάπτυξης, συγγνώμη, και ε, οι στόχοι θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο τα κράτη, αλλά και τους ίδιους τους πρόσφυγες, γιατί και αυτοί έχουν κάποια ευθύνη, θα τους βοηθούμε να επιτυγχάνουν κάποιες λύσεις, να επιτυγχάνουν μια ζωή στα μέρη που πηγαίνουν. Και οι ΜΚΟ φυσικά παίζουν και κάποιο ρόλο στην υποστήριξη του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου. Ε, ξέρουμε ότι η κάθε σύραξη αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή, οπότε οι περιοχές, οι περιφέρειες είναι κάτι που γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει λοιπόν να δοθούν συγκεκριμένοι ρόλοι ε, στους σχετικούς παράγοντες σε κάθε περιοχή. Και τέλος, τα δύο σύμφωνα είναι συμπληρωματικά. Τα σχέδια μηδέν υπάρχουν, έχουν κυκλοφορήσει και για τα δύο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των δύο ε, συμφώνων, διότι πολλά ζητήματα αφορούν και τα δύο σύμφωνα. Αφορούν τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους μετανάστες. Ειδικότερα στο πλαίσιο της, των μεικτών ροών μετανάστευσης ε, ε, σε θέματα όπως είναι η κράτηση, όπως η, βοήθηση, η βοήθεια, η αρρωγή, ε, σε, ευαίσθε, σε ευάλωτες ομάδες, τα παιδιά. Ε, είναι τεράστιο ο κατάλογος. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. γιατί εκπροσωπείται και μη κυβερνητικέ οργανώσει κτλ. Θα προχωρήσουμε τώρα απευθεία στην παρέμβαση του πατρός Φάμπιο Μπατζίο. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας είμαι προσωπικά ευγνώμων ε, που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ιταλικά, γι' αυτό ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φορέσετε ακουστικά, να ακούσετε τους διερμηνείς. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Κλοντ Μωράες, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Βουλίου, γιατί με προσκάλεσε έτσι ώστε να κάνω μια σύντομη παρουσίαση εξ ονόματος της Επιτροπής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες της Αγίας Έδρας, την οποία εκπροσωπώ εδώ. Ε, η σημερινή συνάντηση της Επιτροπής ε, όσον αφορά τους τα παγκόσμια σύμφωνα μου δίνει την ε, δυνατότητα να μεταφέρω την ιδέα που έχει το θέμα αυτό η Αγία Έδρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτική μετανάστευση και ασφαλής μετανάστευσης. Ε, το τμήμα μετανάστευσης, ε, το οποίο ηγείται αυτοπροσώπος ο Πάπας Φραγκίσκος, ε, έχει ολοκληρώσει και εκπονήσει ένα έγγραφο, το οποίο έχει υποβάλει στα Ηνωμένα Έθνη ένα κείμενο 20 τμήματων, 20 σημεία, τα οποία στρέφονται γύρω από τέσσερις λέξεις, υποδοχή, προστασία, προώθηση, ένταξη και αναφέρουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία στο σύνολό τους μπορούν να αποτελέσουν μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση και απάντηση στο θέμα αυτό. Επίσης θεωρήθηκε ε, ε, σκόπιμο να ε, υπάρξει ένα έγγραφο για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα. Επί τη βάσεως της διαπιστώσεως ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες πριν γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλήρη θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της επιλογής αυτής ε, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ευκαιρία που οι διαπραγματεύσεις επί των δύο παγκοσμίων συμφώνων θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο εναρμονισμένες έτσι ώστε να απαντήσουν με τον πλέον προσήκοντα τρόπο ε, εις τις περίπλοκες προκλήσεις της μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης. Στα 20 σημεία αναφέρονται και επιχειρησιακά ζητήματα τα οποία αφορούν ιδιαιτέρως ε, αυτούς που είναι υπεύθυνοι για ε, ε, αυτούς που έχουν αναλάβει την διεθνή προστασία. Πρακτικές οι οποίες προκύπτουν από την επιτόπου εμπειρία των καθολικών εκκλησιών, των Αποστολών και ηρεποστολών. Στοιχείων τα οποία πρέπει να γνωρίζει κανείς η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν βεβαίως ε, να ε, βρουν πολλές καλές πρακτικές ε, στα 20 σημεία του εγγράφου και ακριβώς γι' αυτό το τμήμα μετανάστευσης της Αγίας Έδρας θεωρεί ουσιώδους σημασίας την συνεισφορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν. Οι βασικές αρχές, οι αξίες επί των οποίων βασίζονται τα 20 σημεία δράσης αντιπροσωπεύουν τα πιο, ε, τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία αυτού του ολοκληρωμένου ανθρωπισμού που έχουν σφυριλατήσει διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμφωνίες. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου. Η ανθρωπιστική Ευρώπη, προστάτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, γη ποιητών, φιλοσόφων, καλλιτεχνών, μουσικών, διανοουμένων, μητέρα λαών και εθνών, μητέρα μεγάλων ανδρών και γυναικών, που μπόρεσαν να προστατέψουν και να δώσουν τη ζωή τους για την οξιοπρέπεια των αδερφών τους. Καλείται για μία ακόμα φορά αυτή η Ευρώπη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση. Και εκεί όπου άλλοι αποθαρρύνονται ή λιγοψυχούν, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της δύναμης που τους δίνουν οι παραδόσεις τους μπορούν να ενθαρρύνουν τη διεθνή κοινότητα να απαντήσει από κοινού στις συνολικές προκλήσεις και να εργαστεί για έναν καλύτερο κόσμο ε, στον οποίο ο καθένας θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του η ειδική προστασία ε, στους ετούντες άσυλο και τους ε, πρόσφυγες, ε, τα προγράμματα για τους ανθρώπους αυτούς και οι πολλαπλές νομοθετικές προσπάθειες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, όπως ας πούμε η μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της δέσμευσης που έχει αναλάβει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προβλήματος του ασύλου. Η το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους ε, πρόσφυγες ε, καταδεικνύει ότι θα πρέπει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου αλλά και άλλες Ήπειροι να δεσμευτούν, να στρατευτούν με τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να δοθεί μια κοινή, πιο ευρεία και πιο αποτελεσματική απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα περάσουμε κατευθείαν στην συζήτηση, θα ακούσουμε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας ε, και φαντάζομαι οι πανελίστες θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όλοι σχεδόν στην αίθουσα θέλουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Ε, το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε λίγα λεπτά. Ξέρω πως είστε όλοι οι βουλευτές και θα με λυπηθείτε που πρέπει να προεδρεύσω. Παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε στα δύο λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσω με κάποιον ο οποίος ξέρω τι μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, θα πάμε ευρωβουλευτής, βουλευτής ε, και ούτω καθεξής. Να σε ακούσουμε τους ε, δύο ευρωβουλευτές μας ε, που συνέταξαν την ολιστική προσέγγιση στην ε, μετανάστευση. Ξεκινάμε την κυρία Μετσόλα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Κλοντ. Θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο σύντομη. Η έκθεσή μα βέβαια χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων και σύνταξη οπότε θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα βασικά σημεία. Αλλά Έκτοτε, βεβαίως, ε, το μέγεθος ε, της ε, κατάστασης είναι σχεδόν σουρεαλιστικό, αν μου επιτρέπετε. Ο κόσμος πνίγεται ακόμα, εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν και ως πολιτικοί δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε ότι έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε τα άτομα αυτά να μην είναι απλά στατιστικά στοιχεία χωρίς όνομα. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Όχι άλλες έκτακτες λύσεις για έκτακτες καταστάσεις. Πρέπει να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Και το σημείο αφετηρίας της έκθεσής μας ήταν ότι η ελεγγύη θα πρέπει να είναι η αρχή οποιασδήποτε δράσης για τη μεταναστεύση. Γιατί οποιαδήποτε ολιστική προσέγγιση πρέπει να περιέχει μέτρα τα οποία ως στόχο έχουν πρώτα απ' όλα τα εγκληματικά δίκτυα, τον κόσμο που εκμεταλλεύεται τους πιο αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών που χρειάζονται προστασία και αυτών που έρχονται στην Ευρώπη για να εργαστούν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ενώ αυτοί οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξει έχουν δικαίωμα προστασίας, αυτό δεν σημαίνει κάποιο ε, γενικό δικαίωμα μετανάστευση για όλου πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα της επανακατάστασης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Εάν λοιπόν είμαστε μια ένωση κοινών αξιών, πρέπει τώρα να γίνουμε μια ένωση κοινή ευθύνη. Χρειαζόμαστε ε, βελτιωμένες ασφαλείς και νόμιμες διόδους και μια πιο στιβαρή προσέγγιση στην επανακατάσταση. Αλλιώς, ε, εάν το καταφέρουμε αυτό, ο κόσμος δεν θα μπαίνει σε πιο βαρκές ε, για να πνιγεί. Για την ασφάλεια δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Υπάρχει ε, υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια στους πολίτες μας και τα κράτη πρέπει να πληρούν τις υποχρεώσεις τους στα εξωτερικά σύνορα για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι φόβοι. Μακροπρόθεσμα και τελειώνω. Πρέπει να δούμε τις αιτίε ε, και να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται περισσότερες δεσμεύσεις για να επιλύσουμε τα πολιτικά, γεωπολιτικά ζητήματα της εποχής μας και μια νέα προσέγγιση για την ένταξη που είναι δυτή. Πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων, αλλά λογικό είναι να αναμένουμε και πως όλοι οι άνθρωποι θα σέβονται τις αξίες επί των οποίων ιδρύθηκε η Ένωσή μας. Σας ευχαριστώ, ε, κυρία Μετσόλα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τη Μαλτά. Υπάρχει ένα χορνόμετρο στην οθόνη. Ε, κυρία Μετσόλα, ξεπέρασε τα δύο λεπτά. Παρακαλώ, περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Η κυρία Κιέγγε, σοσιαλδημοκράτης από την Ιταλία, δύο λεπτά. Ε, η κυρία Κιέγγε ήταν ε, συντάκτης μαζί με την κυρία Μετσόλα της σχετικής έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μωράες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους ε, τους ε, καλεσμένους που μίλησαν πριν από μένα ε, γιατί απεικόνισαν και παρουσίασαν πραγματικά όλα τα σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τα παγκόσμια σύμφωνα. Όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρό μας στην αρχή της συνεδρίασης, τα παγκόσμια σύμφωνα αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία λόγω της παγκόσμιας φύσης τους. Αφορούν την κινητικότητα σε όλες τις, τις εκφάνσεις, ε, γιατί είναι συνδεδεμένα τα δύο αυτά παγκόσμια σύμφωνα. Μην λησμονούμε ότι η αποτελεσματική ε, λειτουργία των παγκοσμίων αυτών συμφώνων ε, θα βοηθήσει την κατάσταση να μην είναι πλέον έκθετη. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα σύμφωνα να εφαρμοστούν με τρόπο σωστό και λογικό. Και ακριβώς το μεγάλο θετικό στοιχείο των παγκοσμίων συμφώνων αυτών είναι ότι αφορούν κοινά φαινόμενα και αναφέρονται σε κοινή ανάληψη ευθυνών. Βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης που αποτελεί άλλωστε και το πλαίσιο ε, της ε, ολιστικής προσέγγισης του Κοινοβουλίου μέσω του κειμένου, του ψηφίσματός του, ε, την ολιστική λέω, προσέγγιση των φερμένων αυτών. Ε, είναι θεμελιώδου σημασία να μην λησμονούμε ότι οι χώρες ε, από τις οποίες ξεκινούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει να βοηθηθούν. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκονται στο κέντρο των προσεχών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ακόμα πιο πολύ στο κέντρο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να βρεθούν και αυτά που είπε ο ε, πατήρ Μπιάντζο, δηλαδή ε, τα ε, δικαιώματα, τα ανθρώπινα και άλλα, ανδρών και γυναικών, που υποχρεώνονται να εκτοπιστούν. Η αρχή της μη υποχρεωτικής επανεγκατάστασης, όπως και η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση, θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτά που συνέβησαν στο Μπουρούντι, στο Κονγκό, στην Συρία, τα ανθρώπινα ανθρώπινα σφαγεία όπως τα, έχει αποκαλέσει, τα έχουν αποκαλέσει τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να μην λησμονηθούν. Εάν τα παγκόσμια σύμφωνα καταφέρουν να συνδυάσουν την ρητορική με την πραγματικότητα, θα έχουν κερδίσει πολύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν αυτήν την, και θα χάσουμε όλοι αυτήν την ιστορική ευκαιρία την οποία στην αρχή της συνεδριάσεως ανέφερε ο πρόεδρος Μωράες. Ευχαριστώ. Πάμε στα εθνικά κοινοβουλία. Πάμε στον κύριο Σέγκε Σάλαντ από την Ουγγαρία. Από το ΕΛΚΙ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. If you could uh, put your microphone on, okay, sorry. Is it okay? Just start again. Köszönöm Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρούμε ότι είναι θέμα ισορροπίας, ότι το σχέδιο πέρα από τις υποχρεώσεις θα αναφέρει και τις θεμητές επιφυλάξεις των κρατομελών πέρα από τις ανθρωπιστικές πτυχές πρέπει να έχουμε και τις πτυχές της εθνικής ε, ασφαλείας ε, όταν μιλάμε για την μεταναστευτική κρίση. Συμφωνούμε στο ότι άτομα τα οποία είναι δυνητικά επικίνδυνα θα πρέπει να μπορούν να απελάβνονται άμα τη αφήξη. Χαιρετίζουμε επίσης ε, την σύνδεση με την εξωτερική διάσταση, παραδείγματο χάρη, τις ζώνες διέλευσης και τις ασφαλείς χώρες και είμαστε πεπισμένοι ότι η διαχείριση του προβλήματος πρέπει να ξεκινήσει ήδη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνάψουμε και συμφωνίες ε, όσον αφορά την επανεισδοχή ε, και βεβαίως ε, και όταν μιλάμε για το άσυλο την επανένταξη. Η προστασία των εξωτερικών σύνορων μπορεί να διασφαλιστεί μέσω των hot spot και θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός ε, του τον άσυλο από τους οικονομικούς μετανάστες εμείς. προτείνουμε υπάρξει στο κείμενο η περιγραφή μιας ε, διαδικασίας η οποία θα αναφέρεται στα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται ε, διεθνούς ε, προστασίας και επιπλέον συμφωνούμε να υπάρξουν αποτελεσματικά βήματα στα κράτη εκείνα τα οποία επηρεάζονται περισσότερο για την ένταξη των μεταναστών και για την καταπολέμηση της ε, ρίζοσπαστικοποίησης ε, στις ε, χώρες προέλευσης. Εμείς είμαστε υπέρ της συνεργασίας με των χώρο αυτών. Εμείς δεν θέλουμε ε, πρώτα απ' όλα να υπάρξει μια πολιτική ένταξη θα πρέπει η πρώτη προσπάθεια να είναι η επιστροφή. Ε, Ευχαριστούμε πολύ συναδελφοί ξέρετε αυτά τα δύο λεπτά πρέπει να τα τηρούμε και δεν βλέπω να τα τηρούμε αν μπορείτε παρακαλώ να τα τηρούμε γιατί πρέπει να μιλήσουν όλα τα μέλη και θα πρέπει μετά να έχουμε χρόνο και για την επόμενη συνεδρία. Είναι αδύνατο να συζητήσουμε σε τόσο περιορισμένο χρόνο φυσικά εκτενώ τα ζητήματα αυτά, αλλά όλοι είσαστε, όλοι είσαστε έμπειροι βουλευτές, οπότε είμαι βέβαιο ότι μπορείτε να το επιτύχετε. Η κυρία Ελένη Σταματάκη από το Ιγκούε, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Please go ahead for two minutes, please. Έχετε δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, καθώς οι προβληματισμοί, η ανταλλαγή απόψεων και τα συμπεράσματα της συνάντησής μας θα βοηθήσουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και το σκοπό της ίδιας της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στην τελική διαμόρφωση των δύο παγκόσμιων συμφώνων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και θα γίνουν σεβαστές από το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το 2015, κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη μεγαλύτερη ροή προσφύγων και μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα μιλάμε στη βάση μιας πραγματικότητας που διαμορφώνεται με έναν πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 7 ε, χρόνια στη Συρία, με τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την ασταθή κατάσταση σε πολλές χώρες της Αφρικής, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κρίση που πλήττει τον πλανήτη. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εφαρμόσει πολιτικές που αμβλύνουν αυτή την κατάσταση. Η μόνη μόνιμη λύση στον εκτοπισμό πληθυσμών είναι να σταματήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις, οι ένοπλες σειράξει, οι οικονομικές ανισότητες, η φτώχεια. Το ζήτημα είναι παγκόσμιο και ευρωπαϊκό και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εδωθεί αποσπασματικά είναι απαραίτητη μια κοινή απάντηση η οποία θα στοχεύει και στη ρίζα του προβλήματος, μια κοινή απάντηση που θα προβάλλει την ειρήνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών στη βάση των ιδρυτικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων. Είναι απαραίτητος οπωσδήποτε ένας καταμερισμός ευθυνών ανάμεσα στα κράτη-μέλη που θα διαφυλάσει πρώτα απ' όλα την τήρηση των ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων Παρατηρούνται πάρα πολλές καθυστερήσεις και περιορισμοί στη διαδικασία της οικονομικής επανένωσης των προσφύγων. Σε πάρα πολλά κράτη που αντιβαίνουν τις διατάξεις του Συμφώνου της Γενέβης και του κανονισμού του Δουβλίνου 2, ο οποίος θέτει ανώτατο όριο έξι μηνών για την επανένωση των οικογενειών. Από τις αρχές του 2016, πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης έκλεισαν τα σύνορά τους. ετούντε άσυλο εγκλωβίζονται στις χώρες πρώτης υποδοχής και κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Αυτή η εξέλιξη είχε σαν αποτέλεσμα την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για να μειωθούν οι ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και συνεπακόλουθα προς την Ευρώπη. Η δήλωση αυτή και η συμφωνία είχε πάρα προβλήματα, με βασικότερο ότι αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, το οποίο δεν ισχύει και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που τα αποδεικνύουν. Και είχε ως αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό εγκλωβισμένων ανθρώπων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο υπερπληθυσμός στα ελληνικά νησιά είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ακατάλληλες συνθήκε διαβίωσης που παραβιάζουν βασικά ατομικά ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, Πιστεύω ότι η um, αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη παγκόσμια αντιμετώπιση. Συγγνώμη, μπορώ να σας διακόψω, δεν προλαβαίνουμε. Μεγαλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχή της του Παγκόσμιου Συμφώνου θα πρέπει να είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά... πρέπει να συνεχίσουμε μετά με την επόμενη συνεδρία στις 4 και 4. Αν έχετε άλλο τρόπο, πείτε μου, να μπορώ να το κάνω χωρίς να τηρείτε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έρχεστε και από επιτροπές, ε, όπου και εκεί σίγουρα θα συζητάτε τα πράγματα με περιορισμένο χρόνο. Βλέπω εδώ με κοιτάνε ε, επίμονα μάλιστα, η κυρία Βουέξτρομ με κοιτάει έντονα. Ε, λοιπόν, πείτε μας τα βασικά στοιχεία. Δεν θέλουμε ολόκληρη εκτενώς τη θέση της χώρας σας. Ε, ε, μπορούμε να την δούμε. Λοιπόν, Τερέζα Χιμένες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλόντο. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω το θέμα των διακινητών, δηλαδή ότι οι διακινητές ε, χρησιμοποιούν τελικά την προσφυγική κρίση έτσι ώστε να σπρώξουν τους ανθρώπους ε, στην ε, σκλαβιά. Υπάρχουν δίκτυα διακινητών εγκληματικά. Τα εγκλήματά τους είναι τρομερά, αλλά ακόμα πιο τρομερά είναι τα χρήματα που κερδίζουν μέσα από αυτές στις εγκληματικές διαδικασίες. Άλλο είναι η διακίνηση ας πούμε μεταναστών που σημαίνει ότι βοηθάω μετανάστες ε, να έρθουν για να εργαστούν παράνομα ας πούμε ε, και άλλο είναι το trafficking ε, που είναι στην ουσία το εμπόριο ανθρώπων, η εκμετάλλευση ανθρώπων εντός αυτών των γυναικών και κοριτσιών πολλές προσπαθούν να ζητήσουν άσυλο, αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη διαδικασία διάρκεια της μετακίνησής τους και στη διάρκεια ε, της παραμονής τους σε δομές υποδομής στην Ελλάδα ή αλλού, βιάζονται, αντιμετωπίζουν προβλήματα ε, κλπ. Ξέρουμε ότι αυτές οι γυναίκες, αυτά τα κορίτσια θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν ε, άσυλο γιατί διαφορετικά θα μείνουν στα νύχια των διακινητών. Θα πρέπει να περιγράψουμε σωστά την κατάσταση. Ε, δεν μιλάμε γενικά για θύματα, θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε τις, ε, τα, τα, τα θύματα και θα πρέπει επιτέλους να ποινικοποιηθεί η χρήση ε, των, ε, ε, των διαδικασιών αυτών. Δηλαδή έχουμε ποινικοποιήσει το εμπόριο, το να αγοράσει κανείς στο δρόμο μία τσάντα α πούμε και δεν ποινικοποιείται το εάν κάποιος εκμεταλλεύεται έναν άλλον άνθρωπο. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, δούμε την ε, κατάσταση αυτή όσον αφορά το τράφικινγκ, όσον αφορά το εμπόριο ε, ανθρώπων. Κυρίως πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί τα θύματα είναι πάρα πολλά και η αποκατάστασή τους εξαιρετικά αργή. Από τη Βουλή των Κοινοτήτων, παρακαλώ. Ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ την Επιτροπή μου και υποστηρίζουμε τις αρχές που υπάρχουν σε αυτή την ε, έκθεση. Εμείς ε, για πολλούς αιώνες έχουμε συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Το 1951 παίξαμε σημαντικό ρόλο και είμαστε πρωτοπόροι στην παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης παγκοσμίως. Θέλω να κάνω δύο σχόλια για αυτό το σχέδιο οι πρόσφυγες πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Το πρόγραμμα δράσης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα σχέδια για τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία των προσφύγων. Δεν μπορούν απλά να είναι συμμετέχοντες ε, χωρίς ρόλο. Θέλουμε να γίνει επίσης κάτι για την οικογενειακή επανένωση. Λιγότερη γραφειοκρατία, διεύρυνση του ορισμού της οικογένειας. Ε, υπάρχει μια αναφορά στη σελίδα 13, αλλά είναι σύντομη και ασαφής. Θέλουμε περισσότερο και φυσικά καλωσορίζουμε την παγκόσμια πλατφόρμα, αλλά θέλουμε σαφές χρονοδιάγραμμα και πραγματικό επιμερισμό διεθνώ των ευθυνών. Πρέπει να έχουμε αυστηρά, ισχυρά μέσα με χρονικό περιορισμό. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρξει γλώσσα που να μην μας παρέχει απλά δυνατότητες αλλά υποχρεώσεις και έκφραση βούλησης. Ε, θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, ε, οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε όσον αφορά τα εγγραφά ταυτότητας, ε, οι γυναίκε και τα παιδιά χρειάζονται ασφαλείς χώρους στις τοποθεσίες διεκπαιρέωση προσφυγικών υποθέσεων. Υπάρχουν στα σχέδια κάποιε ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο τολμηρή γλώσσα όσον αφορά τι εναλλακτικέ λύσει αντί για κράτηση ή για κατασκηνώσει να αλλάξουμε το status quo. Αυτό που θέλω να πω εγώ προσωπικά, όποιο και αν είναι η έκβαση του Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνει περισσότερα και όχι λιγότερα και να συνεργάζεται με τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει και κυβερνήσει παγκοσμίω για τον επιμερισμό των ευθυνών τη υποδοχή των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στα έγγραφα με τόση ακρίβεια. Άννα Γκόμες από του ευρωβουλευτέ για του Σοσιαλιστέ. Έχετε δύο λεπτά το πολύ, Άννα. Βεβαίω ε, στηρίζουμε το σύμφωνο, αλλά πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που θα μας βοηθήσει να έχουμε ίσχυη τη συνείδησή μας και δεν θα εφαρμοστεί από τις ε, κυβερνήσεις μας. Ε, έχω βαρεθεί την υποκρισία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και αυτό έχει σχέση και με το κενό μεταξύ της της ε, πράξης και του τι πρέπει να γίνει. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πόσο καιρό περιμένει στο Συμβούλιο αναθεώρηση του Δουβλίνου. Πόσο καιρό ζητάμε να δίνονται ανθρωπιστικές βίζες στους πρόσφυγες. Πόσο καιρό καταγγέλουμε το ότι ευνοούμε τους διακινητές με το να μην ανοίγουμε νόμιμες διόδους για τους πρόσφυγες. Ε, το να πετάμε λεφτά στο πρόβλημα δεν είναι η λύση και να παριστάνουμε ότι κάποιοι άλλοι θα το λύσουν όταν ξέρουμε ότι οι χώρες χώρες δέχονται το μεγαλύτερο βάρος ε, του προβλήματος. Ε, μιλάμε για τη διαδικασία του Χαρτούμ. Όταν στο Χαρτούμ φυλάκισαν ένα, τον Σαλή Μαχμούντο στο Σουδάν που έχει λάβει το βραβείο Ζαχαρόφ, όταν η Αιθιοπία καταραίει με ένα δολοφονικό καθεστώς και δημιουργεί περισσότερους πρόσφυγες ε, και τα ίδια και στην Ερυθρέα. Δηλαδή το να αναθέτουμε σε άλλους η ιδέα ότι μπορούμε να τα αναθέσουμε στη Λιβύη και στην Τουρκία είναι γελία. Επί τη ευκαιρία. Ε, πρέπει και οι εθνικοί βουλευτές να απαιτήσουν λόγοδοσία για το τι συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία που είναι ανήθικη, παράνομη και αναποτελεσματική, όπως είπε και η Ελληνίδα ε, συνάδελφος. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η υποκρισία. Ο κύριος Σάμαν ε, Πεσέτο από το Ελκα από τη Μάλτα για τους εθνικούς βουλευτέ. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I too welcome the, the zero drafts, uh, which I find to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ισορροπία που έχει επιτευχθεί μέσα σε αυτά τα έγγραφα. Βλέπω τα παγκόσμια σύμφωνα ως γενική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, ενισχύσουμε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούν και αλληλεπιδρούν οι χώρες ε, ε, ενώπιον τη τεράστια πρόκληση του ασύλου που όλοι αντιμετωπίζουμε. Θα έλεγα ότι αποτελούν επίση ευκαιρία. μας. δίνουν την ευκαιρία να εμπλέξουμε και να δεσμεύσουμε, ναι, τόσο τι χώρε καταγωγής όσο και τις χώρες διέλευσης στην επινόηση λύσεων που εν τέλει θα μας βοηθήσουν στην υλοποίηση από κοινού. Αλλά εγώ βλέπω τα παγκοσμία σύμφωνα κύριε Πρόεδρε και ως μια δοκιμασία, δοκιμασία δοκιμή των ικανοτήτων μας να μείνουμε ενωμένοι σε ένα ζήτημα το οποίο μέχρι στιγμής έχει αναδείξει ότι υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές μεταξύ μας. Ο επιμερισμός ευθυνών που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, ε, καθώς έρχομαι από μια χώρα στα άκρα της Ευρώπης, τη Μάλτα, είναι μόνο ένα από τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε χωρισμένοι στα Ηνωμένα Έθνη. Ας μετατρέψουμε λοιπόν αυτές τις δοκιμασίες σε μια νέα ευκαιρία. Μια ευκαιρία να μιλήσουμε με μία φωνή σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι στιγμής ε, το ζήτημα των προσφύγων ε, και του ασύλου το βλέπουμε ως πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Και θα μπορούσαν τώρα πλέον, θα μπορούσαν να αποτελήσει όλο αυτό κομμάτι της λύσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να διδραματίσει βασικό ρόλο για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, διότι χρειάζεται αυτή η θέση να είναι σωστή επιτέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, αναγνωρίζουμε το ρόλο σας ε, ως ε, σημαντικό μέλος του Κοινοβουλίου παλιό μέλο του Κοινοβουλίου, ε, κ. Λόπε Αγγιλάρα, ο Ευρωβουλευτής, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα αναφέρω δύο σημεία. Εμείς πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα αντιμετωπίσαμε έγκαιρα τα θέματα αυτά στις κοινοβουλευτικές μας επιτροπές το ζήτημα. Είναι να μην υπάρχει χάσμα ανάμεσα στις αποφάσεις που παίρνουν το, οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εθνικέ συγγνώμη, οι εθνικοί βουλευτές. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση, όπως υπόθηκε εξ αρχής. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τα παγκόσμια σύμφωνα να μην λειτουργήσουν. Τα παγκόσμια σύμφωνα απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, είτε εκπροσωπ εκπροσωπείται η ευρωπαϊκή προσέγγιση από τα ευρωπαϊκά όργανα είτε εκπροσωπείται από εθνικούς εκπροσώπους. Ε, Το, η μετανάστευση, μάλλον ε, να διορθώσω όλοι οι μελητές στα παγκόσμια σύμφωνα για την ε, μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δεσμευτική δρόμη και διάβλη προς την Ευρώπη. Εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Είναι μια σαφής θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εκφραστεί και από το Κοινοβούλιο και από κρατημέλη. Άλλωστε το αποσαφήνισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτική η παροχή ε, ανθρωπιστικών θεωρήσεων, ε, αλλά εάν υπάρχουν τα νομικά μέσα ε, πρέπει οι χώρες να δίνουν την δυνατότητα αυτή. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων να κάνουν ό,τι περνούν από το χέρι τους, ό,τι περνά συγγνώμη από το χέρι τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτές οι νο, αυτοί οι νόμιμοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο κύριος Πέρες Λαπασεράν από το ΕΛΚ και την Ισπανική Γερουσία. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σύντομα θα παρέμβω ως εκπρόσωπος μιας χώρας όπως η Ισπανία που είναι η τρίτη χώρα όσον αφορά την υποδοχή ε, παρατύπων μεταναστών και προσφύγων από τη Βενεζουέλα, από την Κολομβία, από τη Συρία. Σας το λέγω για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε τα θέματα, έχουμε εμπειρία. Θα ήθελα δεν να ασχοληθώ με δύο σημεία τα οποία φαίνονται, αναφέρονται και στη δήλωση του ε, Δουβλίνου και στη δήλωση της Νέας Υόρκης αλλά και σε όποια έγγραφα ε, σχετίζονται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Πρόκειται για αρχές τις οποίες εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικές και αποτελούν ε, ευθύνη των, των κρατών. Ο πατήρ Μπιάντζο το είπε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα κατανοήσουν όλοι. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα φόρουμ κοινοβουλίων και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει αλληλεγγύη να δείξουμε όλοι και ευθύνη να δείξουμε και όλοι και να τη μοιραστούμε όλοι. Πρέπει να επιτευχθεί επιτευχθεί η ισορροπία έτσι ώστε να ε, μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες. Γιατί οποιοδήποτε κανόνας θα σημάνει υπερβολικό βάρος για χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα ή άλλες χώρες οι οποίες δέχονται ε, μεγάλο βάρος προσφύγων και μεταναστών δεν θα λειτουργήσει εάν δημιουργεί, αν προκαλεί αυτό το υπερβολικό βάρος. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονήσουμε στο μέλλον. Ε. Η ευθύνη επίλυσης ε, της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών είναι ευθύνη όλων των χωρών και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα στον κόσμο παντού. Πρέπει να τα λύσουμε όλοι μαζί γιατί διαφορετικά η χιονοστιβάδα των προσφύγων και των μεταναστών δεν θα πάψει να μεγαλώνει. Ευχαριστώ πολύ. Τσάτσεκ το ECR. Szanowni Państwo, e, tak e, wsłuchując się w dzisiejszą Παρακολούθησα την σημερινή συζήτηση ε, και ε, εξακολουθώ να έχω την εντύπωση ότι στην ουσία ε, ε, ε, ε ακριβώς δίνουμε την αντίθετη εικόνα από την Ευρώπη η οποία δεν έχει αλληλεγγύη, η οποία βρίσκεται κλεισμένη από όλε τις πλευρές σε ένα μοναχικό πύργο. Όχι, εγώ βλέπω μια Ευρώπη η οποία εκφράζει την αλληλεγγύη της. Έγινε λόγος για την Πολωνία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο στοιχεία τα οποία έχουν ήδη θυγεί και αναφερθεί. Η εμπειρία της Ουγκάντα, για παράδειγμα, νομίζω ότι θαυμασμό μπορούμε να έχουμε για τη χώρα αυτή, αλλά αναμφισβήτητα θα πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την χώρα αυτή στην προσπάθειά της ε, να ε, δεχτεί τόσους πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες και όχι μονάχα ε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και τη βοήθειά μας αποκλειστικά και μόνο στην Ουγγάντα αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες οι οποίες οι ίδιες έχουν κάνει μια προσπάθεια αλληλεγγύης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, στην κάλυψη των εξόδων αυτών των χωρών οι οποίες είναι γειτονικέ σε χώρες υποσύραξη, οι οποίες ε, προσπαθούν να απορροφήσουν όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό αριθμό προσφύγων. Επίσης, ε, το υφιστάμενο σύστημα ασύλου. Γνωρίζουμε ότι ε, η ε, προστασία των ετούντων άσυλο και των προσφύγων είναι, και των προσφύγων είναι απαραίτητη, είναι διαφυσβήτητη, αλλά θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν η παροχή διεθνούς προστασίας να μειώνει την αίσθηση ασφάλειας της χώρες υποδοχής. Ευχαριστώ από το EFDD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αφαιρθώ στην μορφή της ε, εκδήλωσης η πρόσκληση έλεγε ότι θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ε, κρατών μελών, κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί. Δεύτερον, έχουμε την οπτική εδώ πέρα των παγκοσμίων συμφώνων, τα οποία προσανατολίζονται κυρίως στις ανάγκες ε, των προσφύγων και όχι στην σταθερότητα των ε, χωρών υποδοχής δεδομένων, δεδομένου του αυξανόμενου κόστους ε, που αντιμετωπίζουμε στην ε, χώρα μας, ε, αλλά και ζητήματα εγκληματικότητας και βιασμών ακόμα. Θα ήθελα να τονίσω πως παρά το χτένισμα των επισήμων στατιστικών έχουμε, παραδείγματος χάρη στην δική μου την χώρα, την Βαβαρία, έχουμε σημαντική αύξηση των βιασμών και Βεβαίω, οι πρόσφυγε είναι κατά το 80% που φτάνουν στη Γερμανία νεαροί άντρε. Ε, ταυτόχρονα δεν ε, έχουμε κάποια εμπιστοσύνη στο ότι μπορεί να ε, ρυθμιστεί το πρόβλημα εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο μάλλον να επιληθεί. Γι' αυτό ελπίζουμε στο εθνικό επίπεδο και ακριβώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη πηγή ε, φυγής των ανθρώπων, δηλαδή την κυβέρνηση Μέρκελ. Ευχαριστούμε Μαρτίν Τόλεδαν από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το πρόβλημα του ασύλου, σημαντικό είναι να ξεχωρίσουμε και να μην τον μπερδεύουμε ε, με το πρόβλημα, της, ε, ε, το πρόβλημα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων των μεταναστών με το δικαίωμα στο άσυλο. Δεν είναι δυνατόν πρόσφυγας να θεωρείται κάποιος ο οποίος για οικονομικούς λόγους ή για κλιματικούς λόγους αναγκάζεται να μεταναστεύσει. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, δικαίωμα ασύλου έχει κάποιος ο οποίος ε, είτε υφίσταται, ε, είτε ξεφεύγει, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα πόλεμο, είτε υφίσταται δίωξη για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, φιλής κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο άσυλο. Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη και την παγκόσμια κατάσταση, καλό θα ήταν να κατανοήσουμε τα πράγματα καλά. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε και τον λόγο δίωξης ε, του πρόσφυγα. Γιατί αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα του. Θα πρέπει επίσης ε, να ε, προκύψει μια, ένας μηχανισμός επίλυσης των ενόπλων σειράξεων γιατί ξέρουμε ότι από αυτές τις εμπόλεμες ζώνες φεύγουν οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν άσυλο από εκεί ξεκινούν ε, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη ή αλλού. Και θα πρέπει οι μηχανισμοί να μην αφορούν μονάχα την Ευρώπη και να μην ε, υποδέχεται μονάχα η Ευρώπη πρόσφυγες ε, και δικαιούχους ασύλου, αλλά και άλλες χώρες. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστούν ε, πραγματικά τιμωρία αυτοί οι οποίοι στις χώρες από τις οποίες ξεκινούν οι πρόσφυγες ε, καταπατούν τα δικαιώματά τους και τους φέρνουν σε αυτήν την κατάσταση. Thank you. κάνει από την Νορβηγία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι μέλο του Νορβηγικού Κοινοβουλίου και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μεταξύ σα. Η μετανάστευση είναι ένα φλέγον θέμα παντού και στη δική μου χώρα. Ε, είχαμε εκλογές στο Κοινοβούλιο πέρυσι και το κυριότερο θέμα για την νορβηγική πολιτική ήταν η μετανάστευση. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη ε, μετά από την επίδραση της προσφυγικής κρίσης το 2015. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Το να μην κάνουμε τίποτα δεν είναι επιλογή. Η μετανάστευση θα μας επηρεάσει όλους. Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο των συνόρων πρέπει να συνεργαστούμε. Αν θέλουμε δίκαιο και βιώσιμο σύστημα ασύλου πρέπει να συνεργαστούμε για μια δίκαιη πολιτική επαναπατρισμών και καλύτερη προστασία χρειαζόμαστε περισσότερε πολυμερεί συμφωνίε και χρειαζόμαστε συνεργασία. Και για να κάνουμε κάτι και για τι ριζικέ αιτίε, και εκεί χρειαζόμαστε συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε διαφορετικέ απόψει και το σέβομαι, αλλά το να μείνουμε άπραγοι σημαίνει ότι θα έχουμε σοβαρότατε συνέπειε για όλου μα. Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο σύστημα ασύλου με κοινέ ευθύνε, κοινή πολιτική επαναπατρισμού, ενό συνοριακού ελέγχου. Αυτό χρειαζόμαστε στην ε, Ευρώπη και αυτό αποτελεί κοινή μα ευθύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, ακολουθεί η κυρία Τίτα Φάτνερ από τη Σλοβακία, ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν απαντήσω στο θέμα αυτό να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ίσως ε, ξέρετε ότι χτες οι Σλοβάκοι είχαν μια πολύ θλιβερή ημέρα. Μία δημοσιογράφος, μητέρα δύο παιδιών, ένας δημοσιογράφος, πατέρας δύο παιδιών, ε, δολοφονήθηκε γιατί ερευνούσε κάποιες υποθέσεις διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ελευθερίας ε, του λόγου, γι' αυτό σας διαβεβαιώ ότι η διερεύνηση αυτής της ε, υπόθεσης ε, θα φτάσει μέχρι τέλους στην ε, Σλοβακία και ζητάμε να τιμωρηθεί ο δράστης. Όσον αφορά δε, τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ε, κάποιες προσπάθειες για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ε, πρόσφυγα δηλαδή και οικονομικού μετανάστη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Σλοβακία εδώ και καιρό ζητάει να εστιάσουμε στις αιτίε ε, της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης. Ε, δεν συμφωνούμε να εξάγονται τα προβλήματα αυτών των χωρών. Οι αιτίες ε, της μετανάστευσης πρέπει να επιληθούν εκεί όπου υπάρχουν. Και βεβαίως αυτό αφορά ιδιαιτέρως ε, τις χώρες προέλευσης, τις οποίες δεν μπορούμε να αφήσουμε στην μοίρα του βεβαίως, πρέπει να στηρίξει η διεθνής κοινότητα. Γι' αυτό εκτιμούμε ιδιαιτέρως το ότι στο παγκόσμιο αυτό σύμφωνο υπάρχει μια ξεκάθαρη διατύπωση η οποία απευθύνεται στις χώρες προέλευσης για να αντιμετωπίσουν ακριβώς τα εσωτερικά τους προβλήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού τους. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος από την Λετωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος του Λετωνικού Κοινοβουλίου θεωρώ ότι και τα δύο έγγραφα είναι πολύ ικανοποιητικά. Ήθελα να συγχαρώ και όλους όσους συμμετείχαν στην εκπονήσή τους και όλους τους ομιλητές εδώ. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που μου δίνετε το λόγο, ήθελα να μιλήσω και να μιλήσω κατά των εγκληματικών καθεστώτων που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, το αναφέρομαι στην κυβέρνηση του Κρεμλίνου. Ο δικτάτορας του Κρεμλίνου ε, βάζει τα κρατημέλη να τσακώνονται μεταξύ τους, ε, εξαπατά τους οργανισμούς, τον, Οργανισμό των και αποτελεί τη ρίζα της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Συρία και στην Ουκρανία, καθώς εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε. Έτσι λοιπόν απευθύνω έκκληση προς τους συναδέλφους από τα κράτη-μέλη να τιμωρήσουμε τους Ρώσους υπηκόους που κρύβουν χρήματα στις τράπεζές μας, στέλνουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια και στα σχολεία μας και απολαμβάνουν έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ε, ενώ διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Κάνω έκκληση, όπως και η κυβέρνησή μου, να ε, δείξετε στο Κρεμλίνο ότι δεν μπορεί να καταπατά διεθνείς ε, συμφωνίες ατιμόρυτα. Ωραία. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Ξέρω ότι αυτός δεν είναι ο πιο απλός και καλός τρόπος για να μεταφέρετε τις απόψεις σας. Ε, ωστόσο θα έχουμε κι άλλη μια ευκαιρία ε, να συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και αν δεν είναι η βέλτιστη μεθοδολογία. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις επαφές ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθνικούς βουλευτές που με μετακινήθηκαν, που ήρθαν εδώ, που μίλησαν το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου, τον πατέρα Μπάτζιο, ε, τον ε, αναπληρωτή είπα το εκπρόσωπο ε, και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα, τις παρεμβάσεις τους. Η κυρία Σεσίλια Βίλστρομ θα είναι θα συντονίσει και θα προεδρεύσει αυτή της δεύτερη συνεδρία. Θα προεδρεύσει λοιπόν η κυρία Σεσίλια Βέλστρομ. Είναι και αντίστοιχη συγγήτρια. Δεν θα κάνουμε κανονικό διάλειμμα, απλώς ε, θα χαλαρώσουμε λίγο μέχρι να αλλάξουν θέσεις ε, οι ενδιαφερόμενοι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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και φίλοι. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαίρομαι πάρα πολύ που προεδρεύω αυτού, τη της δεύτερης συνεδρίας για το Σύμφωνο για Ασφαλή Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα με κομψότητα και ηρεμία και ησυχία να εγκαταλείψετε την ε, αίθουσα. Και οι υπόλοιποι να ηρεμήσετε, να, να καθίσετε και να απολαύσετε τη συνέχεια. now we will have the Έλεγα λοιπόν ότι ε, θα έχουμε την ευκαιρία να εργαστούμε με ε, ε, πολλούς υπεύθυνους και ενδιαφερόμενους του θέματος. Πρώτα θα ακούσουμε τους συνδιαμεσολαβητές που θα ηγηθούν των κυβερνητικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων για θέματα σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, δηλαδή τον πρέσβη Χουάν Χωσέ Γκόμε Καμάτσο, μόνιμο αντιπρόσωπο του Μεξικού, καθώ επίσης και τον Γιούρκ Λάουμπερ, πρέσβη ε, και μόνιμο αντιπρόσωπο τη Ελβετία. Πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήρθατε από τόσο μακριά για να είσαστε σήμερα μαζί μας. Το εκτιμούμε αυτό δεόντως. Μετά θα ακούσουμε τον Τζόναθαν Πρέντις, εκπρόσωπο του γραφείου της Λουίζα Άρμπορ. Και μετά τον Εουτζένιο Αμπρόζη, περιφερειακό διευθυντή του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης. Και μετά την κυρία Ιβάντσεβα. Α, δεν είναι εδώ η κυρία Ιβάντσεβα. Τι μου λέτε. Ο κύριος Σιμενόβ όμως είναι εδώ και θα εκπροσωπήσει την, ε, Βουλγαρική Προεδρία και θα μας δώσει μία τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση των πραγμάτων και των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο Συμβουλίου. Τέλος. Θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και βεβαίως ε, πρέπει να ε, πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε και την εκπρόσωπο του Συνδικού ε, Κοινοβουλίου ε, που είναι και συμπατριώτησά μου. Μετά θα είναι η κυρία Μαρία Φέρμ. Μετά θα μιλήσει η Κωνσταντζα Ουρμπάνο Σόουσα, βουλευτή του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας και μετά θα συνεχίσουμε με συζήτηση εκπροσώπων Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά στα πάρουμε με τη σειρά. Θα, θα δίνουμε ε, το, το, λόγο εναλλακτικά όπως και πριν σε ένα, σε ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο Εθνικού Κοινοβουλίου. Εσείς ξέρετε λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνετε, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Υπάρχει ένα έντυπο, μπορείτε να το συμπληρώσετε αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να το δώσετε στη γραμματεία και έτσι θα καταρτιστεί ο κατάλογος των αγορητών. Όμως, ε, ε, από την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν απλώ να ζητήσουν το λόγο ε, και θα του σημειώσουμε. Επίσης, ανάλογα με το πώς οι αγορητέ θα θελήσουν να πάρουν το λόγο, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να περιορίσουμε τον χρόνο αγόρευσης, ο οποίος υπό κανονικέ συνθήκες θα είναι δύο λεπτά. Αφού σας έδωσα λοιπόν όλα τα ε, στοιχεία τα οποία σας είναι απαραίτητα για τα διαδικαστικά, ε, θα ε, δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Μεξικού στον ΟΗΕ, στον κύριο Χουάν Χωσέ Γκόμες Καμάτσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και που μας δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας την άποψη που έχουμε σχετικά με το τι είναι το σύμφωνο ε, ε, για την ασφαλή ε, και ομαλή μετανάστευση. Έχουμε το, zero, το λεγόμενο zero draft, μηδενικό προσχέδιο, το οποίο το σχέδιο 0, ε, επί του οποίου γίνεται η συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά, ε, κυρία Πρόεδρε, ε, που μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την κεντρική πόρτα. Υπάρχει συλλογική συμφωνία των χωρών των Ηνωμένων Εθνών για να διαπραγματευτούμε και να οικοδομήσουμε έναν κοινό τρόπο αντιμετώπισης ε, του μεταναστευτικού φαινομένου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ε, να δημιουργηθεί ε, μία διαδικασία τριών φάσεων. Στην πρώτη φάση όλες οι περιφέρειες, υποπεριφέρειες σε όλο το, από όλο τον κόσμο έπρεπε να κατανοήσουν το φαινόμενο ε, της μετανάστευσης. Ε, εύκολα διαπιστώνει κανείς πόσο λίγα γνωρίζουμε για τη μετανάστευση και επομένως είναι αδύνατον ε, να διαπραγματευτούμε για κάτι το οποίο δεν κατανοούμε. Αυτό κάναμε λοιπόν στην αρχή. Ξεκινήσαμε σε μια πολύ σοβαρή διαδικασία κατανόησης του θέματος αυτό στην πρώτη φάση, αλλά και στην πρώτη και στην δεύτερη φάση το διακύβευμα ήταν να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Να οικοδομηθεί λοιπόν αυτή η εμπιστοσύνη όχι μόνο απέναντι στους δύο ε, συνδιαμεσολαβητές, αλλά και μεταξύ ε, των εμπλεκομένων. Ε, έπρεπε να επιτύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπιστοσύνης ε, που θα μας έδινε την δυνατότητα χωρίς, ε, χωρίς ακραίες τοποθετήσεις να κατανοήσουμε από κοινού κάποια ε, φαινήματα. Είχαμε στην Πόρτο Βαγέρτα στο Μεξικό μια πολύ σημαντική διάσκεψη όπου ε, κατά κάποιο τρόπο ε, εξήγαμε συμπεράσματα σε σχέση με τα όσα είχαν να συζητηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και οι δύο συνεισηγητές, ε, οι συνδιαμεσολαβητές προετοίμασαν το λεγόμενο zero draft. έτσι ώστε να προχωρήσουμε μετά στο Global Compact. Κοιτάξτε, για μα ήταν απολύτως σαφέ ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό είναι ε, μέσω τη συνολική του αντιμετώπισης. Ε, δηλαδή, εάν κατανοήσουμε την μετανάστευση, όχι κατακαιρματισμένη, όχι εστιάζοντας στο ένα ή στο άλλο πρόβλημα, αλλά μέσω μιας συνολικής κατανόησης, να το κατανοήσουμε δηλαδή σαν ένα ενιαίο φαινόμενο. Η προσέγγιση ήταν ε, ε, με προσέγγιση 360 μοιρών. Από την αρχή μέχρι το τέλος πρέπει όλα τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Και νομίζω πως έχετε διαβάσει ήδη το προσχέδιο και θα το ε, διαπιστώσατε φαντάζομαι ότι στο έγγραφο αυτό δεν προωθείται η μετανάστευση, δεν καταδικάζει τη μετανάστευση, αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης. Ε, σε τρία-τέσσερα τμήματα οργανωνόμαστε. Πρώτον, ε, το πρώτο τμήμα αφορά το αφήγημα όχι μόνο του τι σημαίνει Global Compact, όχι μόνο τι περιλαμβάνει και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το Global, Global Compact, αλλά και πώς θα πρέπει ε, να ειδωθεί η μετανάστευση από την πλευρά του Global Compact. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, έπρεπε να ε, σχεδιαστούν και να καταγραφούν 10 βασικές αρχές που θα καθοδηγήσουν την ίδια τη διαπραγμάτευση, αλλά και θα καθοδηγήσουν και την υλοποίηση του Compact, την εφαρμογή του Global Compact. Και επομένως ε, ε, η κάθε αρχή θα έπρεπε να εξηγείται θα βρείτε ας πούμε αρχές όπως είναι τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών ε, να καθορίσουν τις μεταναστευτικές τους πολιτικές, βεβαίως τα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών ε, να καθορίσουν τα σύνορά τους ε, κτλ. Υπάρχουν πολλές πυρηνικές αρχές όπως είναι ας πούμε και το κράτος δικαίου, η δυνατότητα προστασία θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταμερισμός ευθυνών και προσπάθειας κλπ. 22 στόχους έχουμε περιλάβει. 22 στόχους ε, οι οποίοι δεν ε, κατηγοριοποιούνται και δεν περιορίζονται σε κατηγορίες γιατί δεν θέλαμε να κατακαιρματίσουμε την προσέγγιση του φαινομένου την οποία θέλαμε ε, να διατηρήσουμε συνολική και σφαιρική. Ε, απλώς θελήσαμε ε, να δημιουργήσουμε μία αλληλουχία των 22 αυτών σημείων βάσει της αλληλουχίας της μετανάστευσης. Ξεκινήσαμε δηλαδή από την αρχή που είναι ε, η ρίζα του προβλήματος, οι ριζικές αιτίες που οδηγούν στην μετανάστευση, που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν Έλλειψη ανάπτυξης, κλιματική αλλαγή, ε, βίες αλλαγές, ευδία κλπ. Ακολουθήσαμε λοιπόν αυτήν την αλληλουχία, ε, την, ε, την, τον εκτοπισμό, την διέλευση, τα προβλήματα όπως τράφικινγκ και άλλα, μέχρι την άφηξη της κοινωνία υποδοχής. Είναι πάρα πολύ σαφή όλα τα στοιχεία αυτά και οπωσδήποτε είναι προσανατολισμένα προς συγκεκριμένε δράσεις. Η ιδέα του Global Compact είναι να κάνει πραγματικά ασφαλή και ομαλή την μετανάστευση. Το, ε, η επιχειρηματολογία πίσω από, την, ε, από τον σχεδιασμό του Global Compact είναι ότι θα πρέπει να είναι κάτι σαφές ε, και θα είναι προσανατολισμένο στη δράση έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα. Μετά από τους 22 στόχους και τις δράσεις ε, που συνεπάγονται, μας ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη ένας ε, σχεδιασμός για τον τρόπο ε, με τον οποίο ε, και τα Ηνωμένα Έθνη ε, θα πρέπει να κρατήσουν ψηλά στις προτεραιότητες και στις συζητήσεις την υλοποίηση των Global Compact αλλά και τα διακυβεύματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες χώρες. Σημαντικό είναι να πούμε ότι υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν δράσεις, αλλά το Global Compact δεν είναι νομικά δεσμευτικό εργαλείο, είναι όμως ένα εργαλείο το οποίο, του οποίου η υλοποίηση θα βασιστεί ε, στην εμπιστοσύνη και την συνένεση, έτσι όπως αυτή θα διαγραφεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και επομένως είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι δραστηριότητες, στόχοι, δράσεις κλπ ε, δεν είναι ε, ένας ε, υποχρεωτικός κατάλογος, αλλά προτινόμενες δράσεις τις οποίες θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την πραγματικότητα που ισχύει στις χώρες τους, σύμφωνα με το εύρος του μεταναστευτικού φαινομένου, βάσει των ειδικών αναγκών κτλ. Οι ίδιες οι χώρες θα αποφασίσουν ποιες είναι οι πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν. Αυτή είναι μια γενική επισκόπηση ε, των όσων κάναμε και ο συνάδελφός μου ε, ε, Γιώργ Λάουμπερ θα γίνει πιο συγκεκριμένος ενδεχομένως. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Έχουμε άλλον έναν πρέσβη, τον κύριο Γιούρκ Λάουμπερ από την Ελβετία. Είναι πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελβετίας στον ΟΗΕ. Περιμένουμε να σας ακούσουμε κύριε Λάουμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους σας που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Είναι πολύ συναρπαστικά όλα αυτά για μας, διότι φυσικά οι βουλευτές ε, διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία. Οι διαπραγματεύσει μεταξύ των κρατών μελών ουσιαστικά διεξάγονται μέσω διπλωματών, ωστόσο οι βουλευτές ε, αποτελούν ε, το δεσμό με την εγχώρια πολιτική, με τις κοινότητες τις οποίες αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης υπό κάθε μορφή. Η ανταλλαγή αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας και προσβλέπουμε να ακούσουμε όλες σας ερωτήσεις. Θέλω να μιλήσουμε όλοι με μία φωνή, οπότε δεν θα αναλύσω περαιτέρω το σχέδια, αλλά να σας πω εν συντομία πού βρισκόμαστε στη διαδικασία η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά από την υιοθέτηση της διακήρυξης της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 2016. Τα σχέδια που έχουμε αυτή τη στιγμή βασίζονται σε αυτή τη διακήρυξη. Δεν την ε, ε, αναδιατυπώνουν, απλά την πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα. Μέσω αυτού του εγγράφου που είναι πιο αναλυτικό, πιο ακριβές, διαθέτει δράσεις, υλοποίησεις και σχεδιάζει και μια διαδρομή προς το μέλλον για το πώς θα συνεχίσουμε αυτή την παγκόσμια συζήτηση περί αντιμετώπισης της μετανάστευσης. Αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε στη διαπραγματευτική φάση. Έχουμε υποβάλει αυτό το πρώτο σχέδιο στις 5 Φεβρουαρίου. Με ανακούφιση και χαρά δεχτήκαμε πολύ θετικέ αντιδράσει. Οι αντιπροσωπείε θεώρησαν ότι ήταν περιεκτικό το σχέδιο, το αποκάλεσαν ισορροπημένο. Όπω είπε και ο πρέσβη, ανέκθεν ήμασταν πεπισμένοι ότι για να συμμετέχουν όλοι, να συμφωνήσουν όλοι, και να εκπληρώσουμε την εντολή που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη, την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Ε, ε, φαίνεται ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά με αυτό το σχέδιο εγγράφου. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη και από τώρα μέχρι τον Ιούλιο κάθε μήνα θα έχουμε κάποιες λίγες μέρες διαπραγμάτευσης, τρεις-πέντε ε, γύρους θα έχουμε. Μετά από τον πρώτο γύρο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα κρατημέλη διατηρούν τη δέσμευσή τους για το σχέδιο 0, το οποίο όλες χαρακτήρισαν ως πολύτιμο έγγραφο, ως βάση για τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα του που χρειάζεται περαιτέρω εξέλιξη το σχέδιο αυτό. Διάφορα ζητήματα έγιναν πιο σαφή μαζί μας, ως ζητήματα που χρειάζουν περισσότερη συζήτηση με τα κρατη Ο επόμενος γύρος που θα ξεκινήσει λοιπόν σε δύο εβδομάδες ήδη στη Νέα Υόρκη θα είναι αφιερωμένο σε κάποια από αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα από αυτά θα είναι η υλοποίηση, το follow-up και η αναθεώρηση. Σε ποιο βαθμό θέλουν να εμβαθύνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την οικοδόμηση του θεσμικού πλαισίου. και πόσο στο πλαίσιο της υλοποίησης του Παγκόσμιου Συμφώνου θα βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά θα μετατραπούν σε δράση επιτόπου, ώστε η μετανάστευση να αποτελέσει κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής. Αυτά είχα να πω στην παρούσα φάση για τη διαδικασία αυτή. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις της Νέας Υόρκης θεωρούμε ότι οι συζητήσεις για το έγγραφο, για τη μετανάστευση πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό μάλιστα βρισκόμαστε εδώ, για να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με όλα τα θεσμικά οργάνα, με όλα τα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προωθήσουμε αυτέ τι συζητήσει που γίνονται. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από όλου του συμμετέχοντε στην αίθουσα σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη. Ήδη συμπληρώσατε πολύ και εμπλουτίσατε τα όσα μας είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Πάμε στον κύριο Πρέντης. Ε, και στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ε, ξέρετε, στα Ηνωμένα Έθνη εργάζομαι, λέει ο κ. Πρέντε. Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αγαπητό συνάδελφο από το Διεθνή Οργανισμό ε, Μετανάστευσης που κάθεται στα αριστερά μου. Κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας και έχω την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα ζήτημα κορυφαίας Θα Ήθελα επίσης να διαβιβάσω τη χαιρετισμού της Λουίς Αρμπορ, η οποία δυστυχώς ε, κολλείεται σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Κοιτώντας τον τίτλο εδώ πέρα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο και ο ρόλος των κοινοβουλίων, θα ήθελα να προτείνω, αν μου επιτρέπετε, κάποιους τρόπους ε, τους οποίους ε, θα μπορούσατε να σκεφτείτε την σημασία του ρόλου σας στην διαδικασία αυτή στο μέλλον. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση χωρίς υπερβολή είναι μια ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά κάθε γενιά για να εκμεταλλευτούμε τα ωφέλη της μετανάστευσης για όλους τους εμπλεκόμενους και να μειώσουμε τα ε, προβλήματα της. Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης μετανάστευσης τώρα και στο μέλλον, καθώς ε, η δημογραφική, η δυναμική, η περιβαλλοντική και άλλες δυναμικές ε, θα αρχίσουν να αλληλεπιδρούν με τρόπους προβλέψιμους και μη. Στο DNA του συμφώνου, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα τόνιζα τα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά πρώτα απ' όλα την πεποίθηση ότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που θα μας συνοδεύσει για καιρό και για το ότι ο αντίκτυπός της είναι κατά κύριο λόγο θετικός. Δεύτερον, ότι η θετική αυτή πραγματικότητα δεν πρέπει να κρύβει τις πολλές προκλήσεις που μπορεί να έχει η μετανάστευση, ειδικά αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση και κυρίως για τους μετανάστες ίδιους. Τρίτον, ότι για να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της ε, νόμιμης μετανάστευσης ε, και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ε, παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί τη συνεργασία των κρατών. Και τέλος, το Παγκόσμιο αυτό σύμφωνο για νόμιμη ασφαλή και έκτακτη μετανάστευση θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό και της κρατικής κυριαρχίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό εννοούμε εμείς όταν λέμε ότι θέλουμε ένα σύμφωνο το οποίο θα είναι νομικά μη δεσμευτικό αλλά παρόλα αυτά θα εδραιώνεται στο κράτος δικαίου. Ένα σύμφωνο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ε, ανησυχίες των κρατομελών και θα μπορεί έτσι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταναστών και των κοινότητων. Και εδώ είναι ο δικός ο ρόλος Η βουλευτές έχουν έναν μοναδικό ρόλο και κοινοβουλευτικής εποπτείας ε, και ακριβώς ε, τοπικών ανησυχιών και έχουμε έναν ρόλο που σημαίνει προκλήσεις γιατί τα ζητήματα αυτά τα οποία αφορούν την ε, μακροπρόθεσμη ευημερία δεν συμβιβάζονται με τις ανησυχίες της τρέψης πολιτικής. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφέρω τρία σημεία σε σχέση με το σύμφωνο αυτό. Πρώτον, ενώ οποιαδήποτε συζήτηση για, για τα ωφέλη της μετανάστευσης ε, ίσως να βασίζεται μόνο στα γεγονότα, οπωσδήποτε χωρίς τα γεγονότα δεν έχει κάποιο νόημα. Άρα υπάρχει μια ευξενόμενη ανάγκη η συζήτηση για τη μετανάστευση να βασίζεται στα γεγονότα. Γι' αυτό ο στόχος ε, του πρώτου σχεδίου που βλέπετε αφορά ακριβώς τα περισσότερα και καλύτερα και ακριβή και λεπτομερή δεδομένα. Δεύτερον, η ειδική εκπρόσωπος, η κυρία Άρμπορ, έχει ζητήσει προσοχή στο πώς καθορίζουμε την συζήτηση. Βεβαίω ε, δεν μπορούμε να πούμε πως καθοριζουμε την συζητηση βεβαιως όσοι ανησυχούν για τη μετανάστευση είναι ξενοφοβική, δεν μπορούμε να πούμε πως ε, υπάρχει μία σχέση μεταξύ της δημόσιας και της μη ανεκτικότητας. Έτσι περιγράφονται οι μετανάστες ε, είτε παράνομοι είτε οικονομικοί. Έτσι παραγνωρίζεται η ανθρώπινη πλευρά ατόμων που έχουν κάποια ευπάθεια. Και τρίτον έχουμε μία συλλογική ευθύνη να προωθήσουμε, θα έλεγα εγώ, την ένταξη. Αυτό βασίζεται στην έννοια που περιέχει το σύμφωνο αυτό που λέει ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη της ε, μετανάστευσης ε, και για τις χώρες προέλευσης ε, και υποδοχής όπως επίσης ε, και το ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι οφείλουν να εκπροσωπούν και αυτούς οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς και βεβαίω υπάρχει και έννοια του δημοσίου συμφέροντος ε, που εδραιώνεται και στην κυριαρχία που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε ολόκληρες κυριαρχίες ανθρώπων από την προστασία των δημοσίων ε, θεσμών και θεσμικών οργάνων. Κάποια λόγια λοιπόν συμπερασματικά θα ήθελα να τονίσω όπως έκανε και ο βοηθός υπατσαρμοστής για τους προσφύγει, στην παγκόσμια φύση αυτού του εγχειρήματο. Ε, υπάρχει βεβαίω τον τίτλο. Ε, η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τα ωφέλη και οι προκλήσει του δεν περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή και καμία χώρα δεν μπορεί να εφαρμόσει επιτυχώ μια τέτοια πολιτική από μόνη τη. Όταν το αντιληφθούμε αυτό, το πώ δηλαδή οι διαφορετικέ χώρε και οι περιφερειές βλέπουν την μετανάστευση και πώ μπορούν να την αντιμετωπίσουν έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη οποιοδήποτε αποτελέσμα, Η δικιά σα η δουλειά στο διεθνέ ή ε, και στο περιφερειακό επίπεδο όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στόχο να καθυσυχάσει του πολίτε μέσω μια ανοιχτή ε, συζήτηση και η δικιά σα η δουλειά για να στηριχθεί η διαδικασία αυτή θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία έκβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντης και ζητώ συγγνώμη που σας μπέρδεψα με τον κύριο Αμπρόζη. Οφείλεται στο γεγονό ότι στην παρούσα φάση πρέπει κανείς να φοράει τα γαλιά του συνερχώς διαβάζοντας τα χαρτιά που έχει μπροστά του. Θα προσπαθήσω να το συνηθίσω. Λοιπόν κύριε Αμπρόζη, Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια οικογένεια είμαστε, δεν πειράζει πιστεύω, δεν εκνευρίστηκε κανένας, ούτε θύμωσε κανείς με το ε, λάθος, ε, με τη λάθος περιγραφή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε τη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο και χαίρομαι και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ με συναδέλφους και φίλους που μας συνοδεύουν σε αυτή τη συνεδρία. Πολλά υπόθηκαν από τους δύο συνδιαμεσολαβητές και από τον Τζόναθαν ε, για τη διαδικασία για το περιεχόμενο του σχεδίου 0 που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Δεν θέλω λοιπόν να προσθέσω πολλά για αυτές τις πτυχές που ήδη έχουν καλυφθεί. Αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια για τη διαδικασία του Παγκοσμίου Συμφώνου και για τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Θα ξεκινήσω από ένα σχόλιο που έγινε σε μια από τις ερωτήσεις ε, στην προηγούμενη συνεδρία όταν ένας ε, εκπρόσωπος ε, είπε ότι η δράση δεν είναι επιλογή, η μετανάστευση θα μας επηρεάσει όλους. Εγώ θα το άλλαζα λίγο. Θα άλλαζα λίγο αυτή τη δήλωση και θα έλεγα όχι ότι η δράση δεν είναι επιλογή. Θα έλεγα ότι η μετανάστευση θα μας βοηθήσει, θα μας στηρίξει όλους εφόσον πληρούνται μια σειρά συνθήκων και εφόσον πραγματοποιηθούν κάποιες δράσεις. Να σας αναφέρω κάποιες που ήδη ακούσαμε από προηγούμενους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα θα μας υποστηρίξει, θα μας βοηθήσει όλους αν συνεργαστούμε. Αν επιτέλους συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι η μετανάστευση, η διαχείρισή της, η διακυβέρνησή της δεν αποτελούν αποκλειστικά εθνικά ζητήματα. Εξορισμού από τη φύση τους, από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα μετανάστευση από χώρα σε χώρα με τη διέλευση συνόρων αποτελεί διεθνές ζήτημα. Απαιτείται λοιπόν συνεργασία μεταξύ μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία επί ενός κοινού οράματος. Οράματος ε, ε, βέλτιστης διακυβέρνηση του μεταναστευτικού φαινομένου. Κάτι που θα μας βοηθήσει, θα μα στηρίξει όλου για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το κοινό όραμα. Αυτό το κοινό όραμα είναι επίση κάτι απαραίτητο, διότι αντιμετωπίζουμε διάφορες δύσκολε καταστάσεις, διάφορα προβλήματα, προβλήματα συστημικά, όχι προσωρινά, όχι ζητήματα που θα πάψουν να υπάρχουν αύριο, οπότε ε, απαιτείται να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε, να αρχίσουμε να μελετάμε δομικές λύσεις και απαντήσεις, ε, όχι απλά να υιοθετούμε άμεσα προσωρινά, ε, προσωρινές λύσεις. Αυτό είναι το πρώτο εάν. Το δεύτερο εάν, το οποίο θα μα ε, δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη μετανάστευση προ υποστήριξή μα και βοήθειά μα όλων, είναι ότι αν συνεργαστούμε όλοι μαζί προ ένα κοινό όραμα, ε, χωρί να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η διαδικασία, όσα, όλα όσα ακούσαμε να περιγράφονται προηγουμένω, ε, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κατά τύχη, δεν είναι κάτι που μα πέφτει από τον ουρανό βασίζονται σε μια σειρά παλαιότερων δεσμεύσεων της διεθνούς κοινότητας. Η διακήρυξη της Νέας Υόρκης είναι μια τέτοια δέσμευση, η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης είναι μια άλλη δέσμευση. Σε όλα αυτά ε, συνιστάται το επίκεντρο των διαδικασιών όλων αυτών ε, που καταλήγει και στα σχέδια κειμένου που έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά αυτές οι δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλυθεί από την διεθνή κοινότητα πρέπει να συνεχιστούν. Να συνεχίσουν να καθοδηγούν και τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις και την τρέχουσα φάση ε, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γιατί, διότι ε, πρόκειται για δεσμεύσει. Υποτίθεται ότι πρέπει να τις υλοποιήσουμε και να τις τηρούμε. Να τηρούμε τις αρχές που ενέπνευσαν αυτές τις δεσμεύσεις. Και τρίτον, για να, έχουμε, να επιτύχουμε αυτή την υποστήριξη και βοήθεια, αν καταφέρουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία και ελπίζω να καταφέρουμε να τη συνεχίσουμε σε αυτή τη διαπραγματευτική φάση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν αναφερόμαστε σε μετανάστευση, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ανθρώπου. Μιλάμε για πολίτε, του δικού μα πολίτε όλων των χωρών μα, των οποίων εκπρόσωποι βρίσκονται εδώ, των οποίων εκπρόσωποι βρίσκονται στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σε όλο τον κόσμο μιλάμε για ανθρώπου, ανθρώπου με φιλοδοξίε, με δυσκολίε, με όνειρα, με ζωέ, με δικαιώματα. Αυτό το τρίτο στοιχείο Επίσης, πρέπει να είναι παρόν διαρκώς σε όλη τη διαδικασία των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων του Παγκοσμίου Συμφώνου, όπως συνέβη μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι πλέον είναι σαφές ότι αν αυτά οι τρεις συνθήκες που ανέφερα είναι παρούσες στο έργο που έχει επιτελέσει η διεθνής κοινότητα μέχρι στιγμή που εργάστηκε για το Παγκόσμιο Σύμφωνο και είναι σαφές ότι ήταν εκεί. Αντικατοπτρίζονται και αποτυπώνται σαφώς στο ασχέδιο 0 ε, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, οπότε μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί για το πώς ε, είναι η μετανάστευση και η διαχείρισή της η εικόνα μα λέει ότι η μετανάστευση πράγματι θα μα στηρίξει και θα μα βοηθήσει όλου αν τηρήσουμε αυτέ τι δεσμεύσει. Ακόμη δύο λόγια για τα όσα είπε ο Τζόναθαν επίση. Τι ρόλο παίζουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο σε όλα αυτά. Όλοι σα ως εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων και όλα τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου έχετε να παίξετε ένα πολύ σημαντικό τεράστιο ρόλο και βαρύτατη ευθύνη. Πρώτα απ' όλα να διατηρήσετε ε, απαρέγκλητη τη διαδικασία. Εσείς είστε εκπρόσωποι των λαών σας, των λαών της Ευρώπης και έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη διαδικασία θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις, ε, το εγχείρημα αυτό, την προσέγγιση που αποφασίστηκε να υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, ώστε να διασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό αλλά και σε τοπικό επίπεδο ότι αυτός ολικός χαρακτήρας, ε, ολιστικός χαρακτήρας της διακυβέρνησης μετανάστευσης θα είναι μια πραγματικότητα και ότι θα υλοποιείται. Έχετε την ευθύνη να επαγρυπνείτε ώστε να υπάρχει συνοχή πολιτικής, να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι αποφασίζετε από τη μια πλευρά σε σχέση με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της μετανάστευσης να μην έρχεται σε αντίφαση με αποφάσεις άλλων πλευρών, να μην δημιουργούνται παραπάνω προβλήματα σε τομείς πολιτικής ε, σε σύγκριση με άλλους. Και το τρίτο στοιχείο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη δική σας ε, ευθύνη ως βουλευτών είναι ότι ακριβώς επειδή εσείς είστε ο δεσμός μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατικών οργάνων και ανθρώπων και λαών που εκπροσωπείτε, γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει ισχυρή δέσμευση να αλλάξουμε τον τόνο του αφηγήματο τη συζήτηση, κάτι που ακούμε συχνά όσον αφορά τη μετανάστευση. Το αφήγημα αυτό, το οποίο μερικέ φορέ είναι τοξικό, υπερβολικά μάλιστα, που πολύ συχνά δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό στοιχείο και που σε κάποιο βαθμό δεν ε, ε, ταιριάζει και με την ιστορία κάθε χώρας που συμμετέχει εδώ στη συνέλευση αυτήν με το ιστορικό παρελθόν της κάθε χώρας. Οπότε κάνουμε μια προσπάθεια στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του συμφώνου να κρατήσουμε τη μνήμη μας, την ιστορική, να θυμηθούμε τι σημαίνει η μετανάστευση για όλες τις χώρες μας, ανεξαίρετο συγγνώμη από τη δική μου. Μην ξεχνάμε ποτέ από πού ήρθαμε, τι αποτέλεσε η μετανάστευση για μας πώς ε, ήταν μια πραγματικότητα σε διάφορες περιόδους της δικής μας ιστορίας. Ας μην ξεχνάμε αυτή τη μνήμη καθώς αντιμετωπίζουμε όχι την ιστορία αλλά το μέλλον αυτή της διαδικασίας που θα επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αμπρόζη. Ευχαριστούμε που μας θυμίζετε ότι όλοι μας είμαστε μετανάστες από τη φύση μας. Είναι στο DNA μας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά και περνάμε τώρα στον κύριο Σιμεώνοφ που εκπροσωπεί τη Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το Παγκόσμιο Σύμφωνο, αλλά σε αυτήν εδώ την ένωσή μας εσείς είστε οι σημαντικότεροι αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε πάρα πάρα πολλά νομοθετήματα που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε, μελετάμε και πρέπει να ολοκληρώσουμε ώστε να βάλουμε τάξη στα δικά μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μετάξει τη μετανάστευση και να βγούμε από αυτό το χάος το οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε με μεγάλη ανυπομονησία τα σχόλιά σας και να ακούσουμε και για τα εργασίες σας όπως θα εξελιχθούν στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ που καλέσατε και την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Εγώ θα, συμφων... διαφωνούσα ότι ε, βρίσκεται σε χάος η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά ο ρόλος μας ως ε, Προεδρίας είναι πολύπλοκος και δύσκολος. Να βρούμε δηλαδή τον σωστό τρόπο για να οδηγήσουμε το πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατάσταση αυτή αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια συνολική και μακροπρόθεσμη στρατηγική που βασίζεται σε ευθύνη και αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ε, της ε, μετανάστευσης ως ένα παγκόσμιο περιπλοκό φαινόμενο όπως ήδη υπόθηκε που χρειάζεται επίσης παγκόσμιες λύσεις. Ως σημαντικός παράγων ε, στην διεθνή σκηνή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει συνεργασίες για να βρεθούν μακροπρόθεσμες ε, και βιώσιμες λύσεις για την επιτόψη της ε, παράτυπης μετανάστευσης, ενώ έχουμε και νέα μέσα όπως το καταπίστευμα για την Αφρική και οι διάφορες προσπάθειες αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και βεβαίω αυτά μπορεί να μας βοηθήσουν στη μελλοντική διαμορφωσή του συμφώνου. Το μέλλον αυτού του Παγκοσμίου Συμφώνου θα μπορούσε να αποτελέσει την, ε, τον κατάλληλο προσανατολισμό για να μια βιώσιμη και ισορροπημένη προσέγγιση και σε, στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες της μετανάστευσης. Η Προεδρία στηρίζει την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να συνεχίσουν την επικοδομητική τους συμμετοχή στην διαδικασία αυτή, στη Νέα Υόρκη και μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει και στην φάση της διαβούλευσης και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συνεχίσει να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή. Εμεί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα ήταν έτοιμα να μοιραστούν ε, την εμπειρία τους στον τομέα της ε, μετανάστευσης και να χρησιμοποιηθεί για το παγκόσμιο σύμφωνο. Κάποιες από τις βασικές αρχές μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης υπάρχουν, δηλαδή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, η προσοχή ευπάθων ομάδων και η εμπειρία στην διεθνή συνεργασία. Αυτό το οποίο κάνουμε ως Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε ένα συμφωνημένο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το παγκόσμιο σύμφωνο ε, διαπραγματεύσει που γίνονται στη Νέα Υόρκη. Πρώτα απ' όλα θέλουμε ένα ισορροπημένο κείμενο που θα βασίζεται στις αρχές της δήλωσης της Νέας Υόρκης ε, και θα βασίζεται κυρίως στην ατζέντα του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης ε, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι η αρχή της κοινή ευθύνης θα αναφέρεται στις ε, δράσεις ε, του συμφώνου, ειδικά όσον αφορά τις ανάγκες χωρών προέλευσης, διέλευσης ε, και προορισμού και τέλος, να διασφαλίσουμε ότι οι σαφώς καθορισμένοι μηχανισμοί για εφαρμογή και αναθεώρηση θα ακολουθηθούν στα υφιστάμενα φόρα και βεβαίως με ηγετικό ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια, αλλά θεωρούμε ήδη ότι έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο στο τομέα αυτών. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών ε, επεξεργαστούμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και η Σιμιόνοφ. Τώρα η Μαρία Φέρμ ε, θα μας παρουσιάσει την ε, δική της άποψη και ως βουλευτής της Σουηδίας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, η κυρία Φέρμη, οι διερμηνείς δεν ακούν δυστυχώς. Οι διερμηνείς δεν ακούνε αν δεν ανοίξει το μικρόφωνο της η κυρία. Ε, Θα μιλήσω σουηδικά. Βάλτε τα ακουστικά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πάρω το λόγο ε, σε αυτό το ε, φόρουμ. Ε, εγώ θα ήθελα πραγματικά να ε, γίνει λόγος εδώ για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση. Ο τρόπος, με το, το, το πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ε, την μετανάστευση είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι εκτοπισμένοι είναι πάρα πολλοί και όπου η ανάγκη για άσυλο είναι επίσης ε, πάρα πολύ σημαντική. Ε, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε οποιασδήποτε προσπάθειες εμπλοκής και άρνησης του δικαιώματος αυτού. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που πραγματικά χρειάζονται το δικαίωμα στο άσυλο δεν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ε, να οικειοποιηθούν δικαιωμάτων που δεν τους ε, ε, αντιστοιχούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους, άνθρωποι φυσιολογικοί όπως εσείς και εγώ, προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τις διώξεις, από καταστολή ή ακόμα και κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Αναγκάζονται να περάσουν τα σύνορα και αν αρχίζουμε τώρα τώρα να λέμε μα δεν θα έχουν δικαίωμα για άσυλο ε, ή δεν θα έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν του ενός του άλλου δικαιώματος ή ότι υπάρχουν ποσοστώσεις για εκείνο και ποσοστώσεις για το άλλο, τότε οι πιο ευάλωτοι δεν θα έχουν την προστασία που ε, πρέπει και οπωσδήποτε ε, δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που τους αρμόζουν είδαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν ε, σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζουν ε, χιλιάδες συνανθρωποί μας τώρα και επομένως δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να εργαστούμε σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο διεθνές με, με τη βοήθεια των διεθνών συμβάσεων και συνθήκων. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε νέες καταστάσεις. Οφείλουμε να, να, να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι υποχρεωμένοι να φύγουν από περιφέρειες οι οποίες ε, βρίσκονται σε πόλεμο. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε το δικαίωμα στο άσυλο και όχι να το διαλύσουμε. Ε, πολλοί είναι οι λόγοι που οδηγούν ε, τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν. Πολλοί απλώς ψάχνουν μια καλύτερη ζωή, αλλά υπάρχουν και οι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους ε, που φεύγουν από τον πόλεμο. Στην Σουηδία είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε έτσι ώστε να βρούμε ένα σωστό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υποδεχθούμε τους έχοντες ανάγκη θα πρέπει μέσα από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να βελτιώσουν την ε, ζωή τους. Έχουμε όλο και περισσότερους που έρχονται στην ε, Σουηδία που ε, ιστορικά έχει Ε, ιστορικά αποτελεί ε, προσφυλή προορισμό. Ε, το 2015 να σας πω ότι είχαμε 150.000 αιτήσει ασύλου. Είναι γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται θέσεις εργασίας ή έχουμε περισσότερα παιδιά στα, σχολεία, στα σουηδικά σχολεία. Ωστόσο αυτό δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από από μια αλληλέγγυα η υποδοχή και θα πρέπει βεβαίως να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες και προϋποθέσεις υποδοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πρωτίστως δε στις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και όμως όλες αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν ε, με ε, συμμετοχή της ε, Ευρώπης. Θα πρέπει να είναι σαφής η νομική κατάσταση, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οποιασδήποτε φες ζώνες. Η εγκατάσταση και η μετεγκατάσταση ξέρουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε καταστάσεις όπου λόγω ποσοστώσεων δεν θα γίνονται ε, δεκτεί κάποιοι άνθρωποι και δεν θα ε, εφαρμόζεται η αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε συνανθρώπους μας στα χέρια των διακινητών και δεν μπορούμε να αφήσουμε ανθρώπους να διακινδυνεύουν τη ζωή τους ε, καθημερινά. Γιατί διαφορετικά ο αριθμός των θυμάτων διαρκώς θα αυξάνεται. Στην ε, Σουηδία ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση ε, έτσι ώστε να μελετήσουμε τα σημεία ε, επί των οποίων μπορεί να υπάρξει βελτίωση του συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν ε, ασφαλείς ε, διαβλή για την μετανάστευση μέσα ας πούμε από ανθρωπιστικές θεωρήσεις, βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους δηλαδή, μέσα από την ε, έκδοση ε, ε, μικρής διάρκειας αδειών παραμονής κλπ. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το βράχι πρόθεσμο και να προχωρήσουμε προς το μάκρο πρόθεσμο που είναι η παροχή ασύλου σε, στους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που το χρειάζονται. Ε, ε, επίσης μπορούν να υπάρξουν και άλλοι λόγοι όπως είναι σπουδές, ανώτερες σπουδές ή μεταπτυχιακά, ε, οικογενειακή επανένωση. Το, ήδη στην Σουηδία έχουμε ένα σύστημα ιδιαίτερα ανοιχτό όσον αφορά τους εργάτες και γενικά το εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Είναι γεγονός ότι βλέπουμε πολλούς που δουλεύουν ε, χωρίς άδεια που δουλεύουν στη μαύρη αγορά. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε. Ε, ε, μέσα στους πρόσφυγες μπορεί κανείς να βρει άτομα με προσόντα, με ικανότητες τις οποίες η σουηδική αγορά χρειάζεται. Το σημαντικό είναι να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στην νόμιμη αγορά εργασίας. Ε, είδαμε ποιες ε, είναι οι ανάγκες ε, σε ειδικά προσόντα και προσπαθήσαμε να τις καλύψουμε και μέσα από τους πρόσφυγες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται ε, την διεθνή προστασία αλλά δεν καταφέρνουν να την ε, επιτύχουν. Ξέρουμε ε, και βλέπουμε όλοι καθημερινά τα ατυχήματα αλλά και τις εγκληματικέ ενέργειες και τις δολοφονίες κατά των μεταναστών στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά, κυρίως δε τα παιδιά που έρχονται μόνα τους στην Ευρώπη, οι ασυνόδευτοι ανήλικες είναι ανήλικες, ανήλικες συγγνώμη, είναι ε, πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, πρόβλημα ε, και δεν μας ενδιαφέρει γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στις χώρες μας, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Και στρέφομαι τώρα, λέει η Προεδρεύουσα, στην κυρία Κωνσταντζα Ουρμπάνοντε Σόουσα, που εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Έχετε το λόγο, αγαπητή κυρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, υπογράψω, να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα αυτής εδώ της ε, συνεδρίασης ε, μετά από την επιτυχία του Παγκόσμιου Συμφώνου που δεν θα είναι δεσμευτικό νομικό, νομικά οπότε η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των κρατών ε, και το πόσο καλόπιστα θα δράσουν οι χώρες. Μιλήσαμε για μετανάστευση εδώ εκτενώς. Ωστόσο δεν έχουμε ορίσει το πλαίσιο σωστά, διότι η διεθνής μετανάστευση σήμερα είναι εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Μην ξεχνάμε ότι μόνο το 3,5% σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα είναι πληθυσμός μεταναστών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν φεύγουν από τη χώρα τους, από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι. Ανέκαθεν υπήρχε μετανάστευση, είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Περίπου η ίδια ήταν η ένταση. Είναι σίγουρα είναι πιο περίπλοκο το φαινόμενο της μετανάστευσης σήμερα, πιο διαφοροποιημένο, πιο πολύμορφο, αλλά υπάρχουν αλλαγές ε, όπως υπάρχουν αλλαγές στα πάντα. Ε, πρέπει αλλά, έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουμε τη μετανάστευση αποφασιστικά. Αντί να βλέπει κανείς τη μετανάστευση θετικά, ο κόσμος αρχίζει να αποκτά αίμονες ιδέες, θεωρώντας τη μετανάστευση ως μια απειλή. Εδώ και περίπου 20 χρόνια θεωρείται συνδεδεμένη με την παρανομία, το έγκλημα, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα. Έτσι χαρακτηρίζει τη μετανάστευση. Και αυτό αξιοποιείται από τι λαϊκιστικέ μάζε, κάποια λαϊκιστικά ρεύματα που παίζουν με του φόβου των ανθρώπων, του εκμεταλλεύονται για να ε, διαστρεβλώνουν την μετανάστευση, διαστρεβλώντα την εικόνα τη ενώ πρόκειται για κάτι φυσικό, κάτι απαραίτητο και θετικό, Όπω υπήρξε πάντα για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο το σύμφωνο αυτό, αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο, μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία μοναδική, ώστε επιτέλους να δοθεί τέλος στο ανθρώπινο, στην ανθρώπινη τραγωδία που είναι σήμερα η ανθρώπινη μετανάστευση, να κοπεί επιτέλους αυτός ο φαύλος κύκλος που συνδέει την παρανομία, τα περιοριστικά μέτρα, όλο και μεγαλύτερη παρατυπία και παρανομία, γόνιμο έδαφος για τις εγκληματικές οργανώσεις και που δυσκολεύει τα κράτη-μέλη στη διαχείριση του φαινομένου αυτού. Είναι μια μοναδική ε, ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της παγκοσμιοποίησης. Αν ε, δούμε καθαρά την παγκοσμιοποίηση, χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση, αυξημένη, την απελε... αυξημένη απελευθέρωση των κινήσεων, της κυκλοφορίας, των εμπορευμάτων, ε, των ανθρώπων, των υπηρεσιών, αλλά δεν χαρακτηρίζει αυξημένη κυκλοφορία των ανθρώπων. Η λογική δηλαδή που διακατέχει όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα, την κυκλοφορία κεφαλαίων και ανθρώπων και, και εμπορευμάτων συγγνώμη, και υπηρεσιών, δεν χαρακτηρίζεται την κυκλοφορία των ανθρώπων, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ε, ε, το αντικείμενο εθνικής, ε, εθνικών ρυθμίσεων περιοριστικών, που βασίζονται σε μια λογική περιορισμού, απαγόρευσης διατήρησης ε, της εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους. Είναι το τελευταίο κομμάτι εθνικής κυριαρχίας που έχει απομείνει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο να βασιστεί στην αποδοχή ότι δεν θα καταφέρουμε ποτέ να καταλαγιάσουμε αυτό τον άνεμο, για να το πω κάπως ποιοτικά, της, ε, της μετασταναστευτικής κίνησης, ούτε με τους ελέγχους στα σύνορα, για να καταπολεμήσουμε τη μετανάστευση πρέπει συλλογικά να διαχειριστούμε το φαινόμενο αυτό και θεωρώ ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Για το σχέδιο 0 θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε ξανά και ξανά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εργασιών. Τι διακρίνει έναν δικό μας πολίτη από έναν ξένο, ένα σύνορο. Σιγά, σήμερα είμαι πολίτης μιας χώρας και αύριο γίνομαι μετανάστης, δεν πάω να είμαι άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την εικόνα θα πρέπει η μετανάστευση να γίνεται κατανοητή με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη και να θεωρούμε τη μετανάστευση ως κάτι φυσικό και μάλιστα ουσιαστική σημασία για την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Οι στόχοι του συμφώνου είναι πολύ αριθμοί βέβαια, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στο λίγο χρόνο που μου απομένει σε τέσσερις. Στην ε, καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων εμπορίας ε, ανθρώπων, αυτή ε, η μάχη πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το επόμενο σημείο. Ο έλεγχος των συνόρων και οι ποινικέ διώξεις κατά αυτών των δικτύων είναι απαραίτητα μέτρα μεν, ωστόσο δεν πρόκειται ποτέ να είναι αρκετά για να δώσουμε τέλος σε, αυτή την τραγωδία. Το δεύτερο, δεύτερο μέτρο, μόνο χάρη στη δημιουργία βέβαιων, ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης. Θα καταφέρουμε να έχουμε στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε την απώλεια ανθρώπινων ζωών, διότι επειδή ακριβώ λείπουν αυτές οι νόμιμες οδοί, οθούμε ανθρώπους στα εγκληματικά δίκτυα που λειτουργούν όλο και πιο περίπλοκα, ε, αποκομίζοντας όλο και μεγαλύτερα κέρδη καθιστώντας τον κόσμο μας ένα κόσμο αποτρόπαιο που εκμεταλλεύεται εσχρά τις ελπίδες των άλλων. Πρόκειται για μια αγορά που λειτουργεί βάσει της αρχής της προσφοράς και της ζήτησης. Και επίσης ε, θα πρέπει να παρέμβουμε ώστε οι χώρες και κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες να καταλάβουν πολύ καλά ότι η πραγματική κρίση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μες στην επόμενη δεκαετία δεν θα είναι μεταναστευτική αλλά το δημογραφικό, η δημογραφική κρίση. Να γνωρίζετε ότι η μείωση του πληθυσμού και η γύρανση του πληθυσμού θα θέσουν πιέσεις στην οικονομική μας ε, ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα των κοινωνικών μας συστημάτων. Γι' αυτό το λόγο η μετανάστευση αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση μια άριστη ευκαιρία για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την οικονομική μας πρόοδο, τη βιωσιμότητά της και η νόμιμη μετανάστευση θα αποτελέσει μια ουσιαστική οδό που θα διασφαλίσει, θα εξασφαλίσει την ασφαλειά μας. Γιατί δεν είναι η μετανάστευση που δημιουργεί την αβεβαιότητα, αλλά τα εγκληματικά δίκτυα, οι εγκληματικοί οργανισμοί που εμείς στηρίζουμε, που εμείς τροφοδοτούμε, που αποτελούν απειλή κατά της δικής μας ασφάλειας. Στη συνέχεια υπάρχει επένδυση στις πολιτικές ένταξεις, είναι το τρίτο απαραίτητο μέτρο. Η μετανάστευση, όπως είναι φυσικό, επιφέρει αλλαγέ στις κοινωνίες και όπως όλα τα φαινόμενα μετασχηματισμού, μεταλλαγής και ανάπτυξης ε, προκαλεί δυσκολίες. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αποτελεσματικά πολιτικά μέτρα ένταξης τα οποία δεν θα αφορούν μόνο τους ανθρώπους που υποδεχόμαστε, αλλά θα αφορούν και τις κοινωνίες υποδοχής, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε αυτές τις κοινωνίες υποδοχής, οι οποίες πρόκειται να μεταλλαχθούν, να αλλάξουν ε, μέσω θρησκευτικών εντάσεων, ε, ε, εθνοτικών τάσεων ή άλλων εντάσεων. Και τέλος, δεν θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε όλους τους μετανάστες του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε και ένα ανθρώπινο δικαίωμα που είναι το, ανθρώπινο, το δικαίωμα να παραμείνει κανείς στο σπίτι του. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τις δομικές αιτίες που οδηγούν στη μετανάστευση. Ώστε η μετανάστευση να είναι μια επιλογή και όχι πλέον μια υποχρέωση. Μια προενεργή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να συνοδεύεται πάντα από σοβαρές πολιτικές καταπολέμησης των ε, αιτιών της μετανάστευσης. και που, αιτίες που δεν έχουν αλλάξει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο πόλεμος, η ανασφάλεια, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η πείνα, η φτώχεια. Αυτό σπρώχνει τους ανθρώπους ε, στη μετανάστευση. Αυτές είναι οι βαθιές αιτίες της μετανάστευσης, όχι οι δικές μας πολιτικές, ούτε η εξωτερική μας πολιτική. Ε, πρέπει να δεσμευτούμε σοβαρά στην πρόληψη των ένοπλων σειράξεων, να επενδύσουμε στις ε, πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας οι οποίες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές πρέπει να αλλάξουμε και τις δικές μας εσωτερικές πολιτικές την κοινή γεωργική πολιτική για παράδειγμα ή την εμπορική μας πολιτική ώστε να δώσουμε και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μια πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης δημιουργώντας συνθήκες τέτοιες που θα δώσουν τη δυνατότητα βελτίωσης της ζωής αυτών των πληθυσμών. Ένα πράγμα είναι βέβαιο ε, αν βασιζόμαστε στους έλεγχους στα σύνορα, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ε, στη ε, εξωτερικό έλεγχο των συνόρων, όλες αυτές οι πολιτικές θα είναι αναποτελεσματικές ε, για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης με βέβαιο τρόπο. όσο θα υπάρχει μια σοβαρή προοπτική καλύτερη ζωής αλλού, οι άνθρωποι αυτοί θα μετακινούνται και θα είναι αδύνατον να τους σταματήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ και εγώ κυρία Ουρμπάνο Ντεσόουζα και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για τις ε, παρεμβάσεις σας ε, που πραγματικά μας συγκίνησαν. Τώρα θα δώσω λόγο στους συναδέλφους και να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε με την κυρία Βαλενσιάνο από την Ισπανία, Ευρωβουλευτή. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σημειώσω πόσο σημαντική είναι αυτή η συνάντηση, γιατί η παρουσία εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων, η συνεργασία <clears throat> με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, εάν θέλουμε πραγματικά ε, να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο ε, σύμφωνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, άσκησε επανειλημμένα κριτική ε, όχι τόσο στην ενωσιακή όσο σε εθνικές πολιτικές για την μετανάστευση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και σωστό και δίκαιο να υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων. Το είπαν σχεδόν όλοι οι παρεμβαίνοντες. Νομίζω ότι ε, η κατάσταση είναι κρίσιμη και θα είναι αποφασιστική σημασία για τα επόμενα χρόνια το θέμα αυτό. Ενδεχομένως το ζήτημα της ε, μετανάστευσης ε, μα, δημιουργεί πρόβλημα και προκαλεί σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, ε, των ακραίων ε, εκδηλώσεων σε πολλές ε, χώρες και είναι γεγονός ότι πολλές ακραίες πολιτικές ομάδες και σχηματισμοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευαισθησία. Ο λαϊκισμός σιγά σιγά όμως δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και σε εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, που, πολιτικών κομμάτων που είναι αντίθετοι προς τέτοιες κινήσεις όπως και φαινόμενα όπως ε, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε μια ευρεία οπτική γωνία και να δούμε πώς θα συνεχίσει η Ευρώπη ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση, ε, η προσφυγιά δεν είναι φαινόμενα τα οποία θα σταματήσουν αύριο. Και θα πρέπει πραγματικά να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ε, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, θα ήθελα να μάθω εάν θα υπάρξει κάποιο έγγραφο κοινό το οποίο θα υποβληθεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, ε, προτίθεται το Συμβούλιο να οικοδομήσει, ας πούμε, να διαμορφώσει ε, μια ευρωπαϊκή θέση παρά τις όποιε διαφορές. Δεύτερον, εάν υπάρχει ένας μηχανισμός υλοποίησης για αυτό το σύμφωνο ή εάν το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και θα ήθελα να σας πω ότι την 5η Απριλίου παρελθόντος έτους ε, ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για, την, ε, για τον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Το ψήφισμα είχε συγγραφεί από την κυρία Βαλενζιάνο και από τον κύριο, ε, και από τον κύριο Ντίας Ντεμέρα. Πραγματικά σας συστήνω να διαβάσετε το έγγραφο αυτό, είναι πολύ ε, ε, καλό. Το εγκρίναμε την προηγούμενη χρονιά και καλή για συντονισμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ελένη Σταματάκη από την Ελλάδα. Παρακαλώ αυτή τη φορά όμως να μην ξεπεράσετε το χρόνο σας, δύο λεπτά το πολύ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Μια παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή τακτική και κανονική μετανάστευση θα πρέπει να εστιάσουμε στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού του στάτους και στα ωφέλη που μπορεί να έχουν τα κράτη από την πολιτισμικότητα. Να σεβαστούμε τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως επιτάσσει το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και να διασφαλίσουμε την προστασία από φαινόμενα διακρίσεων και ρατσισμού. Να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπη και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στη δικαιοσύνη, να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη γλώσσα τους, να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους έφηβους, για τις γυναίκες, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να παρέχουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και να τους δώσουμε πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Ε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της τεράστιας οικονομικής κρίσης και του τεράστιου προσφυγικού κύματος, εφαρμόζεται ένα πολύ πετυχημένο σχέδιο για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Έχει νομοθετηθεί από το 2016 η δυνατότητα μεταναστών χωρίς χαρτιά να δουλεύουν νόμιμα με εργόσιμο. Έχουμε διευκολύνει τη διαδικασία έκδοσης αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ετούντες άσυλο ώστε να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έχουμε, εξετάζουμε την νομοθετική ρύθμιση για πρόσκοπη εγγραφή των προσφύγων και μεταναστών στα Μητρώα Ανέργων και στην ένταξή τους σε προγράμματα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι κάποια μέτρα στα οποία νομίζουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την νόμιμη ε, ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες μας ε, στην προσπάθεια αυτή έχουμε στήριξη από τα κινήματα αλληλεγγύης και από την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον τρόπο αυτό ε, ε, πιστεύουμε ότι η ένταξη θα είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πήρα λίγο χρόνο παραπάνω, με συγχωρείτε. Αλλά... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Now I turn to Mr. Perez Lapa. Στρέφομαι τώρα στον κύριο Πέρες Λαπασαράν από την Ισπανία, από, από την Ισπανική Γερουσία, από το ΕΛΚ. Κύριος Λαπαθαράν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος ε, χώρας ε, της Ισπανίας, θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι παγκόσμιες συμφωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πιστεύουμε επίσης ότι η μετανάστευση όντως πρέπει να είναι ασφαλής, ομαλή και τακτική, αλλά θα ήθελα να υποβάλω και κάποια ζητήματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι σημαντικά, σημαντικές. Ναι, πρέπει να βελτιώσουμε βεβαίω τη μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να εξαρτάται αυτό από την εξωτερική πολιτική. εξωτερική πολιτική ε, των δυνάμεων, των χωρών, των κρατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, μεγαλύτερη συνεργασία. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε συνεργασία γίνεται από μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει οπωσδήποτε ως βασικό στοιχείο να περιλαμβάνει και την συνεργασία για θέματα ε, μεταναστευτικά. Υπάρχουν χώρες της ε, Αφρικής ε, που όμως δεν, με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε αν έχουν υπάρξει συμφωνίες ή όχι. Εμείς στην Ισπανία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα, στις πόλεις οι οποίες είναι κοντά στα σύνορα και στα σύνορά μας γενικότερα. Θέλουμε να δημιουργηθούν καλές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, ε, κοινέ ερευνητικές ε, μονάδες, ε, κοινά προγράμματα. Τέλος, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτό κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Eurojust, η Europol και οι υπηρεσίες εγκληματικών ερευνών εθνικές και διεθνείς θα πρέπει οπωσδήποτε να, να, έχουν ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε μετανάστευση θα γίνει πραγματικά ασφαλής και ομαλή. Ε, θέλ, ε, πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να δεχτούμε μετανάστες αλλά στις χώρες μας, αλλά οπωσδήποτε να ελέγχεται ταυτόχρονα ε, και το μεταναστευτικό ρεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφός μου, κύριος Λόπες Αγγιγιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για όλους τους πανελίστες ε, αναφέρετε το, αυτό που θα πω, γιατί πραγματικά ε, τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Η μετανάστευση είναι συνδεδεμένη και με την ανθρώπινη φύση. Αλλά αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα δεν είναι μονάχα μια μεταναστευτική κρίση η οποία σε λίγο θα περάσει. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, ευρωπαϊκή απάντηση, τρόπο διαχείρισης, αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στο προηγούμενο πάνελ είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση ανάμεσα ε, στα δύο θέματα το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη μετανάστευση θα πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά για να μπορέσουμε εν τέλει και στο παραδεχτούμε να αλλάξουμε αυτό το αρνητικό πρόσημο που είχε πάντα η ευρωπαϊκή προσέγγιση τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών. Κοιτάξτε, ε, οι άνθρωποι κάνουν, ε, γίνονται παράτυποι μετανάστες γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι νόμιμοι μετανάστες. Εάν θέλει κανείς να βρεθεί εδώ, θα πρέπει να γίνει παράτυπος μετανάστες, ε, μετανάστης ε, και μάλιστα πολλές φορές με τρόπους ε, που τον αναγκάζουν να γίνει και παράνομος μετανάστης, όχι απλώς παράτυπος. Επομένως θα πρέπει επιτέλους να ανοίξουν νόμιμες οδοί έτσι ώστε να μπορέσει η εθνική νομοθεσία να ε, δώσει τουλάχιστον ε, θεωρήσεις, ε, βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και τίποτα. Κυρία Πρόεδρε και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρτιν Τολεδάνο. Δεν μας είπε η Πρόεδρος από πού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Por España, del Congreso Και εγώ από την Ισπανία είμαι, αλλά όχι από τη Γερουσία, από τη Βουλή. Κοιτάξτε, εδώ αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσουμε, να διαρθρώσουμε μια ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση. Μια νόμιμη μετανάστευση δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι Μία τέτοια μετανάστευση μπορεί να είναι θετική, γιατί το μέλλον των χωρών μας, λόγω ακριβώς της, της δημογραφικής κρίσης, ε, προϋποθέτει και παρουσία άλλων ανθρώπων, παρουσία μεταναστών. Και επομένως αυτό το δέχεται θετικά και η κοινωνία. Και εμείς πάντα θα είμαστε απέναντι στον λαϊκισμό ε, σε αυτόν που διώκει τον ξένο, τον μετανάστη, έτσι ώστε να αναπτύξει πολύ αρνητικές πολιτικές. Πιστεύω ότι η αλληλεγγύη ε, θα πρέπει να είναι κύριο, ε, κύριο γνώρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσει μέσω αλληλεγγύης και τις χώρες εισόδου όπως είναι η Ισπανία, όχι μονάχα τις τελικές χώρες υποδοχής για, τους, ε, για τα παράτυπα κύματα μετανάστευσης θα πρέπει να ε, δημιουργηθεί ένα σωστό σύστημα ε, καταμερισμού έτσι ώστε πραγματικά να είμαστε δίκαιοι γιατί εμείς στην Ισπανία είμαστε σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρα χρειαζόμαστε επίδειξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης από ό,τι άλλες χώρες. Θα πρέπει να δουλέψουμε επίσης ε, και στις ε, χώρες ε, προέλευσης, χώρες οι οποίες λόγω της οικονομικής τους κατάστασης προκαλούν τη μετανάστευση των πολιτών τους. Θα πρέπει να γίνουν συμφωνίες ανάπτυξης αλλά και συμφωνίες επιστροφής στις χώρες προέλευσης των παρατύπων μεταναστών. Και επίσης ε, θα πρέπει να ποινικοποιηθούν όλες οι δράσεις και κινήσεις αυτών ε, των εγκληματικών οργανώσεων ε, οι οποίες κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί είναι μαφίες αυτές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση ως εκπρόσωπος της ε, Γερμανικής Βουλής. Η μετανάστευση είναι ένα παγκοσμίο πρόβλημα και βεβαίως αυτονόητο είναι το ότι χαιρετίζουμε το ότι και ο ΙΕ ασχολείται με το θέμα και προσπαθούμε να αναζητήσουμε από κοινού μια λύση στο πρόβλημα. Θα ήθελα εδώ πέρα να σας διαβεβαιώσω ευκαιρίας δοθήσεις ότι η Γερμανία είναι οπωσδήποτε αξιόπιστος ε, εταίρος στην συζήτηση αυτή για να βρεθεί μια λύση τους επόμενους μήνες και χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2015, έχουμε αποδείξει πως ε, έχουμε μεγάλη, μεγάλο ανθρωπισμό και αλληλεγγύη. Βεβαίως αυτό οδήγησε και σε αρνητικές συνέπειες στον πολιτικό διάλογο στην χώρα μας και είπε ο κύριος Πρέντς ότι πρέπει να είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί στην συζήτηση. Συχνά βλέπουμε και ξενοφοβία ε, και στα κοινοβουλιά μας. Γι' αυτό εμείς θέλουμε ειδικά σε θέματα ασύλου και προσφύγων, να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι για εμάς στο Τσεντεού Τσεσού αυτό έχει ε, μεγάλη σημασία, δηλαδή να συνεχιστεί η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thanks to you. Χάρη και σε εσά λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κυρία Γκόμες. Ε, με κάλυψε η κυρία Κωνσταντ Ουρμπάν Σόζα να πω πως ήταν ε, και υπουργό εσωτερικών. Συμμετείχε στη συζήτηση και ξέρει τι λέει όταν λέει ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον αέρα με τα χέρια μας, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη μετανάστευση με ελέγχους. Ε, το θέμα είναι η διαχείριση ε, από κοινού. Και τώρα να το δούμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και να το επικοινωνήσουμε θετικά, γιατί χρειάζεται η μετανάστευση, γιατί έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Ένωση και ωφελούμαστε από αυτήν. Και το θέμα είναι να μην συνεχίσουμε να ταΐζουμε τα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών που εκμεταλλεύονται το ότι δεν έχουμε νόμιμες και ασφαλείς διόδους είτε για πρόσφυγες είτε για μεταναστές και επί τη ευκαιρία έχουμε νόμιμα συστήματα. Τα περισσότερα μάλιστα είναι εκτός ελέγχου και εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου από τα Εθνικά Κοινοβούλια να δουν το τι συμβαίνει με τα συστήματα αυτά, τα λεγόμενα χρυσή βίζα, προγράμματα επενδυτών μέσω των οποίων κινδυνεύει η ασφάλεια του συστήματος Σέγγεν και εκπορνεύουν την υπηκότητά μας στα άτομα αυτά που είναι πλούσια και παριστάνουν ότι είναι παγκόσμιοι πολίτες. Δεν θέμε τέτοια σκουπίδια και διαφθορά. Αυτά είναι ξέπλυμα χρήματος, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να διαχειριστούμε τη μετανάστευση για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις ζωές τους εργαζόμενοι και συνεισφέροντας στις κοινωνίες μας. Αυτό χρειαζόμαστε και πρέπει να γίνει συλλογικά και όχι με τις χρυσές βίζες. Δεν θα υπηρεστούμε έτσι τις κοινωνίες μας. Wow, finally we have... Επιτέλους, ε, ακούω κάποιες αντιδράσεις από την αίθουσα. Κύριε Σέγγερ Ζάλν από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω και να προειδήσω ότι σε, αυτήν, σε αυτό το σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και λοιπά μετανάστευση ε, αναφερόμαστε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγες και οι οποίοι δεν καλύπτονται από την ε, Συνθήκη της Γενέβης. Η παρούσα κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη και πολλές χώρες έχουν, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω των μεταναστών. Στην Ουγγαρία δεν ε, μπορώ να πω ότι ε, συμφωνούμε ε, με, το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Εντάξει, δίνονται κάποια θετικά παραδείγματα και με αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, απ' την άλλη μεριά όμως δεν είναι δυνατόν να ε, δεχτούμε και τους οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι απλώς έρχονται στην Ευρώπη για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ούτε είναι δυνατόν ε, να ζητήσουμε από μια άλλη χώρα να βοηθήσει κάποια χώρα η οποία έχει πάρα πολλούς μετανάστες. Υπάρχουν ε, φυσικά εμπόδια, υπάρχουν θεσμικά εμπόδια ε, στις διαδικασίες. Ε, γίνεται λόγος για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση. Αν θέλουμε την οικονομική μετανάστευση, την μετανάστευση για οικονομικούς λόγους, να την εντάξουμε σε ένα τέτοιο σύμφωνο, ε, τότε τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθε χώρα μέλος θα πρέπει ε, ανεξάρτητα και κυρίαρχα να παίρνει τις αποφάσεις του. Ευχαριστώ. one final request for the floor. Νομίζω ότι έχω ένα τελευταίο αίτημα για να πάρει το μικρόφωνο κάποιος. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εντίτα Φούντνερ από τη Σλοβακία. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να μιλήσω αρχικά, αλλά ακούγοντας αυτή τη συζήτηση πήρε μια τέτοια τροπή που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. μιλάμε για ευρωπαϊκά συστήματα τα οποία να λειτουργούν και ξαφνικά ακούω αντιδράσεις και εγώ εκ μέρους της Σλοβακίας ε, έχω να σας πω ότι η Σλοβακία μπορεί να χειριστεί τις ελλείψεις στην αγορά εργασία της μέσω της μετανάστευσης αλλά θέλουμε να επιλέγουμε από ποιες χώρες θα λαμβάνουμε οικονομικού οικονομικούς μετανάστες στη, και θα του εντάσσουμε στο εργατικό μας δυναμικό είναι χώρε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από τη Σερβία. Γιατί αλλιώ η μετανάστευση, ξέρετε, αναδεικνύει διαφορέ θρησκευτικέ και άλλε διαφορέ ε, μεταξύ των εθνών μα. Το ταξίδι στο οποίο έχουν επιβαστεί κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το επιβάλλουν σε άλλα κράτη δεν μπορούν να υποχρεώσουν κάποια κράτη να υποδεχθούν υποχρεωτικά κάποιον αριθμό μεταναστών προσφύγων. Αυτά τα συζητάμε και βάσει πραγματικών εμπειριών και μου κάνει έκπληξη η αντίδραση κάποιων ανώτατων Ευρωπαίων πολιτικών που απειλούν ορισμένε ε, χώρε ότι θα τι αποκλείσουν ε, από την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψη Αποφάσεων απλά επειδή σκέφτηκαν να έχουν μια διαφορετική άποψη για την επίλυση αυτού του προβλήματο. Θέλουμε να συμμετέχουμε, αλλά με διαφορετική άποψη, διαφορετικέ μεθόδου για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και μα κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη που κάποιε χώρε όπω η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία ε, θα συμμετέχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι ευρωπαϊκά κράτη για λογαριασμό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ούτως ή άλλως μας απειλούν. Ευχαριστούμε, ήσασταν απόλυτα σαφείς. Μάλιστα, σαφές ότι υπάρχουν και εντάσεις ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Ευρώπη όταν μιλάμε για μετανάστευση. Παρ' όλα αυτά έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες και προκλήσεις ε, πολύ μεγαλύτερες από αυτήν. Είμαστε μια πολύ τυχερή περιοχή του κόσμου με 28 κράτη-μέλη, ε, προσεχώς 27. Παρ' όλα αυτά, 500 εκατομμύρια άνθρωποι με το υψηλότερο στο αλφαβητισμού, με το χαμηλότερο στο παιδικής θνησιμότητας, ε, έχουμε τόσα πολλά πράγματα που πάλι άνθρωποι στον πλανήτη μόνο όταν ονειρεύονται μπορούν. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε μέρος της λύσης όταν μιλάμε για το παγκόσμιο αυτό σύμφωνο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ασφαλή, έφτακτη μετανάστευση, για διαχείριση της μετανάστευσης και θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και να το υπομισθούμε από κοινού. Όπως είπε κάποιος από τους πανελίστες, καμία χώρα δεν μπορεί να το διαχειριστεί από μόνη της. Αλλά μαζί μπορούμε να είμαστε ισχυροί και να το διαχειριστούμε από κοινό. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είδαμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών και ε, συναδέλφων από διάφορες ε, χώρες. Ελπίζω λοιπόν να επιτύχουμε μια καλύτερη αντίληψη και μεγαλύτερο σεβασμό Με αυτές τις παρατηρήσεις λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πάνελ αυτό και ευχαριστώ θα δώσω την Προεδρία στην συνάδελφο την κυρία Σουίτσα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε καθίστε για να περάσουμε στη τελευταία ε, φάση της συνεδρίασης ε, και να κλείσουμε. Είναι όλοι κουρασμένοι πλέον, ας προσπαθήσουμε να κλείσουμε. Στα γρήγορα παρακαλώ καθίστε. Thank uh, Σας ευχαριστώ όλους. Όπως ξέρετε, ερχόμαστε στο τελευταίο τμήμα της σημερινής ε, συνεδρίασης. Πριν κλείσουμε με τα συμπεράσματα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκ Τζακομίνη. που εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Πρέση Εξωτερικής Δράσης Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε κρίσιμη στιγμή αμέσως μετά την παρουσίαση του Παγκοσμίου Συμφώνου και του Σχεδίου 0. Χαιρόμαστε που έχει το έγγραφο αυτό και το θέμα αυτό να την προσοχή του Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε που συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβουλία στη συζήτηση. Και στη συζήτηση αυτή εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και με την υποστήριξη των Εθνικών Κοινοβουλίων θα δημιουργήσουμε τα δύο σύμφωνα αυτά. Η μετανάστευση είναι παγκόσμιο ζήτημα. Η διακήρυξη της Νέας Υόρκης αποτελεί ορόσημο ανάδειξής της ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βασικές αρχές ε, που θεσπίζονται εκεί είναι η αλληλεγγύη, η επιμερισμένη ευθύνη, η δέσμευση και παραμένουν αυτές κατευθυντήρες αρχές. Ε, ανοίγουν το δρόμο προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο αντιμετώπισης της μετανάστευσης ως παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως είπαν πολλοί ομιλητές σήμερα, πάνω από 65 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται παγκοσμίω ως πρόσφυγες, ε, ετούντες άσυλο οι μετανάστες. 258 εκατομμύρια διεθνεί μετανάστες υπάρχουν παγκοσμίω, οι περισσότεροι από του οποίου εργάζονται και ταξιδεύουν τακτικά. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος συμμετέχων έχει οικοδομήσει μια ολοκληρωμένη μακροχρόνια στρατηγική βάση ελληνικής και, ε, και συνεργασίας. Σώζει ζωές και προστατεύει τις ζωές ε, ε, προσφύγων και μεταναστών, καταπολεμά την εμπορία ανθρώπων και δημιουργεί νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη. γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης των ριζικών αιτιών της μετανάστευσης και του αναγκαστικού εκτοπισμού με νέα εργαλεία όπως τα Trust Fund, όπως τη Βαλέτα, που επικεντρώνονται στους νέους και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ε, μέσω αυτών των νέων προσεγγίσεων ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις πρακτικές και τις εμπειρίες ε, ε, για την αντιμετώπιση των νέων ζητημάτων. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο περιθώριο. Χρειάζεται να συμμετέχουμε όλοι στις ε, λύσεις, χώρες καταγωγής, χώρες προορισμού, χώρες διέλευσης. Όλες μπορούν να υποφεληθούν από τη διεθνή συνεργασία. Το πρώτο κομμάτι της συζήτησης αφιερώθηκε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση για τους πρόσφυγες, συγγνώμη. Υποστηρίζουμε την UNHCR στο σημαντικό εγχείρημα ανάπτυξης ε, των ε, ολοκληρωμένων αποκρίσεων με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες. Όπως ανέφεραν και άλλοι ομιλητές, η αλληλεγγύη βελτιώνει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και είναι κρίσιμη σημασία. Ο επιμερισμός ευθυνών η συμμετοχή όλων των κοινωνιών και ο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους πρόσφυγες. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε ισορροπημένη ε, συμφωνία, ισορροπημένο σύμφωνο που να καλύπτει και τις προσδοκίες των χωρών και απαλύνοντας τις πιέσεις προς αυτές. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, Χαιρόμαστε που ακούσαμε τις απόψεις των πρέσβεων Καπότσο και Λάμπερ ε, για την διακυβερνητική διαδικασία. Ήταν άριστο επίτευγμα αυτή η δημιουργία του εγγράφου του σχεδίου 0 που αποτελεί βάση για τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα πλήρες έγγραφο, ισορροπημένο, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Με γνώμονα τον βασικό σκοπό της ασφαλούς ε, ε, τακτικής ε, ομαλής μετανάστευσης. Χαιρόμαστε για αυτή την προσέγγιση που είναι επικεντρωμένη σε ανθρώπους, ειδικότερα όσον αφορά ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση, ειδικότερα τα παιδιά. Και λαμβάνοντας υπόψη και τη διάσταση του φύλου. Επίση, χαιρόμαστε που δίνετε προσοχή στην αναπτυξιακή διάσταση και χαιρόμαστε που έγινε πρόταση για συγκεκριμένες δράσεις ώστε να καταπολεμήσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο των εμπόρων ανθρώπων. Θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσει για να διευκρινίσουμε καλύτερα τα διάφορα ζητήματα που περιέχονται στο σύμφωνο, όπω ενίσχυση τη συνεργασία για την αντιμετώπιση τη άτυπη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών υποχρεώσεων διευκόλυνση του επαναπατρισμού ή τη επανεισδοχής μέσω μια προσέγγιση, βασισμένη στον άνθρωπο, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε των μεταναστών μαζί με τον σεβασμό των αξιών, των ανησυχιών και των αναγκών των κοινωνιών, των χωρών καταγωγής και των χωρών προορισμού. Εδώ εξετάζουμε ζητήματα όπως ε, ένταξη, δυνατότητα απορρόφησης των αγορών εργασίας ε, κτλ. Και τέλος συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε έναν βασικό ρόλο ε, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε θέματα υλοποίησης στο, πλαίσιο, στο ευρύτερο πλαίσιο των Ηνωμένων η συνεργασία, η δέσμευση αποτελούν αρχές για μας. Η πρόσφατη δημιουργία μιας Task Force ε, Ηνωμένων Εθνών Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της, κατάστασης, της ανθρωπιστικής κατάστασης της Λιβύης, στη Λιβύη αποτελεί υπόδειγμα των όσων μπορούμε να επιτύχουμε μαζί με τους εταίρους μας στον τομέα της μετανάστευσης. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή στην όλη συζήτηση. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, το όλο εγχείρημα και τη Βουλγαρική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε να τηρούμε ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουμε την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Ολομέλεια το Μάρτιο. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας. Ευχαριστούμε και θα σας στείλουμε ενήμερους ε, για τα αποτελέσματα και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τον κύριο Κλοντ Μωράς, για τις τελικές του... Τα τελικά... Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Ήταν ε, πολύ μεγάλη ημέρα, θα ήθελα να φέρω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εθνικούς βουλευτές, ειδικά όσους έμειναν μέχρι το τέλος. Η διαδικασία αυτή είναι μία από τις πιο ευαίσθητες, ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα για τα εθνικά κοινοβούλια. Το γνωρίζουμε αυτό. Γνωρίζουμε πως υπάρχει ένα φάσμα απόψεων εντό των κρατών μελών που τις ακούσαμε σήμερα. Γνωρίζουμε επίση πως υπάρχουν κράτη-μέλη που βρισκόνται σε διαφορετική κατάσταση ε, και στην φορτικά κομμάτια της παγκόσμιας κρίσης. Μιλάμε για την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Γερμανία. Ακούσαμε από την Πορτογαλία κάποιες χώρες ε, Βίζεγκραντ. Το θέμα είναι ότι τα γνωρίζουμε αυτά γιατί και οι βουλευτές μας είναι από αυτές τις χώρες ε, και νομοθετούν. Οπότε τα γνωρίζουμε αυτά. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε τις αιτίες της μετανάστευσης ε, από συγκεκριμένες ε, χώρες. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο σύμφωνο, δύο παγκόσμια σύμφωνα που διαχειριζόμαστε τώρα και πρέπει να εμπλακούμε για τα θεσμικά όργανα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Συμβούλιο, για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για την Κομισιόν, από την οποία ακούσαμε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συνομοθέτης, γύρω στο 40% της ε, νομοθεσίας ε, της ε, Προεδρίας αυτής αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε επαφή και να πούμε κάτι για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία ήταν λοιπόν η σημερινή, παρά το ότι γίνεται με τρόπο δύσκολο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συνέβη. Δεύτερον, πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τρίτον, τι κάνουμε τώρα. Το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα θα καταλήξουν σε ένα ψήφισμα τον Μάρτιο, όσο το είναι τον πιο ισορροπημένο. Ε, η Λίμπε, η οποία κάνει το νομοθετικό κομμάτι και αναφέρθηκαν κάποια από τα ζητήματα, θα πάμε τον Δεκέμβριο στο Μαρόκο και θα οργανώσουμε περισσότερες ε, συνεδριάσεις για το Παγκόσμιο Σύμφωνο και θα εργαστούμε με τρόπο ολιστικό και Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα έχει μια ανταλλαγή απόψε, 25 Απριλίου και θα εργαστούμε όλοι για να έχουμε μια συνεκτική διαδικασία και τέλος να πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα σε πολλά κράτη-μέλη και εδώ. Οπότε η σημερινή συνεδρίαση δεν έλυσε όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά εκτιμούμε το ότι ήρθατε εδώ και συνεισφέρετε στην διαδικασία αυτήν. Είναι καλύτερο να μπλακούμε σε αυτήν την διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μην έχουμε εμπλακεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συμμετοχή σας και οπωσδήποτε έμαθα πολλά σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, μπορείτε να ολοκληρώσετε τώρα την ε, συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Μωραές, ευχαριστώ Κλοντ για τις παρατηρήσεις σας αυτές, για τα καλά σας ε, λόγια, για το έργο της Επιτροπής ε, Λίμπε, η οποία είναι η Επιτροπή στην οποία υπάρχει το περισσότερο νομοθετικό έργο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ πως η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο λόγω της σημασίας του Παγκόσμιου Συμφώνου, αλλά επειδή τα κράτη-μέλη ακριβώς ε, οδηγούν αυτές τις ε, διακρατικές διαπραγματεύσεις. Τώρα γνωρίζουμε πως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο σε όλες τις ε, χώρες μας. Όπως ακούσαμε, χρειάζεται μια ευρωπαϊκή ηγεσία, άρα η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη και πρέπει να έχουμε ένα κοινό όραμα. Καμία χώρα, όπως ακούσαμε σήμερα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα μόνη της. Η συνάντηση αυτή είχε στόχο ακριβώς να έχουμε ένα κοινό όραμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τους επόμενους μήνες ε, και θα δούμε και τι θα γίνει με την έγκριση του συμφώνου που προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Τα κοινοβούλια πρέπει να ακουστούν σε αυτήν την συζήτηση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό της μετανάστευση και του εκτοπισμού. Πρέπει να εμπλακούμε κι εμείς ε, θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας σε αυτήν την συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές ε, που ήρθαν σε αυτήν την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση για τις εξαιρετικές τους συνεισφορές. Σας ευχαριστώ λοιπόν και καλό σας βράδυ.